Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας και παρακαλώ όλους σας στις θέσεις σας για το θέμα της σημερίσιας διάταξης θα ήθελα να σας κάνω αρκετά σχόλια. Επειδή έχουμε πολλά θέματα, η κυρία Τσίμερη, η συγγήτρια, μας λέει ότι θα υπάρξει εξέταση των συμβαστικών ε, τροπολογιών στην έκθεσή της για τις συνέπειες της κρίσης ακριβώς ε, και για τις ίσες ευκαιρίες ανάμεσα άνδρες και γυναίκες. Είναι το σημείο 6, αλλά θα έχουμε αύριο την ψηφοφορία. Η συγγήτρια και πάλι, Σταϊνρίκ για το σιδογνωμοδότησης για τις ε, Στο σημείο 20 θα αλλάξει το σημείο αυτό και θα γίνει το 16α. Και με τη συγκίτρια συμφωνήσαμε ότι το 19 για τις τροπολογίες για την έκθεση κ. Καζάς, για την έκθεση της Επιτροπής, για την οδηγία για νέες εταιρικέ σχέση για τις υπηρεσίες. Ε, στο σημείο 19 αυτό αναβάλλεται για μια άλλη συνάντηση. Είναι το σημείο 21 τώρα που θα πρέπει να εξετάσουμε για τον κύριο Μπουλάν για ε, σύσταση σώματος για ανθρωπιστική βοήθεια. Θα το εξετάσουμε σήμερα το πρωί και θα αποτελέσει το σημείο 13α. Και επίσης ε, για την κατάσταση για τους συντονιστές, για την πρόταση της Επιτροπής ε, για τις υπηρεσίες ακριβώς. Έκθεση ΜΑΝ ε, και εργαζόμαστε με την Επιτροπή Μεταφορών. Προσθέθηκε το σημείο αυτό σήμερα το πρωί και θα είναι το 21α. Και για τις συνάντηση των συντονιστών να σας πω κάτι. Η ψηφοφορία για την έκθεση του κ. Σόγκορ δημογραφικές στατιστικές στο σημείο 29 αυτό αναβάλλεται για άλλη συνάντησή μας. Εντάξει, τώρα περνάμε στο σημείο 2, αν έχετε κάτι να προσθέσετε εσείς, είναι οι ανακοινώσει της Πρόεδρου σας. Μετά από τη συνάντησή μας ε, θα γιορτάσουμε ανάμεσα στα μέλη ακριβώς ε, της Επιτροπής μας ε, την καινούργια χρονιά και θα είμαστε σίγουροι περισσότεροι εδώ. Και ακόμα κάτι, γιατί είχαμε ζητήσει από την Νομική Επιτροπή για τη έτοιμά μας στο δικαστήριο και έχει επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελευταία της πρόταση σχετικά με το ΡΕΣ. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων λοιπόν ασπάστηκε την άποψή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσφύγει για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τρίτη ανακοίνωση, τόση γνωμοδότηση του Στίβεν Hughes για την Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων. Έκθεση της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων ε, θα την έχουμε μόνο μέσα Φεβρουαρίου. Γι' αυτό οι τροπολογίες ε, για το θέμα αυτό που είχαν προβλεφθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου ισχύουν τώρα μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου το μεσημέρι ώστε να λάβουν υπόψη τους ε, την ε, έκθεση Πεντεμπισεύκο όταν ακριβώς θα την έχουμε. Και ακόμα κάτι να σας υπενθυμίσω ότι η διακίνηση η κοινοβουλευτική αυτή εβδομάδα έχει μεγάλη σημασία. από τη Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, 28 με 30 Ιανουαρίου και έχει ε, ιδιαίτερα σπουδαίο ρόλο να παίξει η Επιτροπή μας με την Επιτροπή Νοτιματικών Υποθέσεων και Προπολογισμού και παρακαλώ να είστε παρόντες όσο γίνεται περισσότεροι και στη συνάντησή μας ε, την Τρίτη το απόγευμα που εμείς θα καθοδηγούμε ακριβώς θα έχουμε την απασχόληση των νέων και τα διάφορα σχέδια για την λιτότητα. Και μέσω του δικτύου ναι, αναμεταδίδεται η συνάντησή μας. Τώρα ο συνάδελφός μας Στέφεν Χιούζ έχει το λόγο για την έξαση των συμβαστικών τροπολογιών, για την έκθεσή του, για τους κινδύνους λόγω του αμοιάντου στην ε, υγεία, στην εργασία και οι προοπτικές ε, αφαίρεσης αμοιάντου εκεί που υπάρχει ακόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους και εισηγητές και τους υπόλοιπους βουλευτές που συνεργάστηκαν στενά μαζί μου για το θέμα αυτό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Ζορτ Μπακ σκιώδη εισηγητή από άλλες ομάδες. Εργαστήκαμε εδώ για να ετοιμάσουμε για να ετοιμάσουμε πολλές τροπολογίες ταυτόχρονα Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε τα πρόσθετα σχόλια των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων συναδέλφων και βεβαίως θα διευκρινιστούν περαιτέρω οι τροπολογίες. Δεν θα τις ε, διατρέξω. Είχαν την ευκαιρία οι συνάδελφοι να τις διαβάσουν πιστεύω. Δύο από τις σημαντικότερες, η GKH για την G Εδώ θέλουμε να δούμε τι δυνατότητε δημιουργία ενό προγράμματο για την απομάκρυνση του αμοιάντου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μελέτη αντικτύπου και την ε, διασταυρούμενη, την πολλαπλή ανάλυση. Την ανάλυση τη πολλαπλή συμμόρφωση. Βλέποντα το παράδειγμα τη Πολωνία με τι δυνατότητε απομάκρυνση ε, του αμοιάντου στο 2032. Η καθοριστική τροπολογία, κατά την άποψή μου, είναι εκείνη που συστήνει τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μητρώα, καταλόγους δηλαδή για την, καταγραφή του, για την καταγραφή του αμοιάντου και να διοργανωθεί σωστά η εξάλληψη του αμοιάντου. Κυρίως για να προστατευτούν και εργαζόμενοι που μπορεί να εκτίθενται σε κινδύνους από την ουσία αυτή τα μελλοντικά χρόνια. Αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες αντικαθιστούν κάποιες από αυτές που αρχικά είχαν υποβληθεί. Υπάρχουν κάποιες κοινές τροπολογίες με την κυρία Μωράν Σαρτιά και τον κύριο Μπακ. Ελπίζω και αυτές να υποστηριχθούν. Απλώς δεν μπορώ να στηρίξω τις, τις τροπολογίες της κυρίας Ασέα. Με σκοπό σχεδόν να εξαλείψουν την έκθεση, το μεγαλύτερο μέρος της τουλάχιστον. Όμως θα συμφωνήσω με πολλές από τις ε, ε, τροπολογίες του κυρίου Μπακ και της κυρίας Τζανόνη. Um, the final point... Και του κυρίου Λουκά. Επίσης, Κάτι που επεσήμανε ο κύριος Κλάρκ στην περασμένη συζήτηση. Ήθελα να ξέρω, να ξέρω ότι συμμερίζομαι μέρος των επιχειρημάτων του. Το θέμα του Λευκού Μιάντου και το κατά πόσον ενέχει σημαντικούς κινδύνους ήταν κάτι για το οποίο υποσχέθηκα στους συναδέλφους πληροφορίες. Επεσήμανα ότι το έχει καταγράψει ως επικίνδυνη ουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύπτεται και από το πρόγραμμα REACH. Και πραγματικά χθε λάβαμε μια πολύ καλή ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι μπόρεσαν να το κοιτάξουν. Το καλύτερο θα ήταν να μοιραστεί εδώ στην αφήσα τη Επιτροπή. Την περασμένη φορά δεν πρόλαβα να τα παρουσιάσω στην Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι είναι καρκίνογόνο επικίνδυνη ουσία κατά την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής η ουσία αυτή. Η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να γίνει πριν από 15 και 20 χρόνια, όταν συζητούσαμε ακόμη αν θα απαγορευτεί ο αμύαντος γενικότερα. Πρόεδρε, θα περιμένω να ακούσω τις απόψεις των υπόλοιπων συναδελφών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρτήρια στον εισηγητή μας, τον Στέφεν Χιούζ, γιατί συνεργάζεται πολύ καλά όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Χαίρομαι γιατί τα θέματα της υγείας ε, λόγω του αμοιόντου, δεν χαίρομαι μάλλον, γιατί δεν φαίνονται καθαρά τα προβλήματα του αμοιάντου και παραμένουν είτε σε πλοία, είτε σε δημόσια κτίρια, σε σύραγγες κλπ. Χαίρομαι όμως ε, για την ε, συμφωνία μας ε, ώστε για το θέμα αυτό και το ότι οι εργαζόμενοι δυστυχώς όμως από την άλλη μεριά δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει κυρίως σε θέματα κατασκευών, συντήρηση κλπ. και δεν γνωρίζουν καθόλου την παρουσία μιάντου. Γι' αυτό η έκθεση αυτή θα πρέπει όλα τούτα να τα δείξει καθαρά. Και χαίρομαι γιατί συμφωνούμε να πούμε στην Επιτροπή να κάνει μια σύσταση στα κράτη-μέλη για δημόσια μητρώα, για δημόσια αρχή, καταγραφή ακριβώς εκεί που βρίσκονται ακόμα αμύαντος και να ενισχύσουμε την προστασία του κόσμου και να ενισχύσουμε την προστασία του στον χώρο εργασίας και θα πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει σε σύσταση μιας εργασία ε, που να έχει σχέση με την αμίαντο και τα επαγγέλματα εκείνα που αφορούνται ιδιαίτερα όπως όσοι εργάζονται σε σε κατασκευές ε, κλπ. Και έχουμε το λάμδα το λατινικό, την συμβαστική λύση που ζητάμε μια οδηγία που να καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής κατάρτισης ακριβώς για όλους που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς και εκεί όπου επεξεργάζονται τα απόβλητα αμοιάντου. Αυτά είναι τα θετικά σημεία που ήθελα να πω μέχρι τώρα, εκεί που συμφωνήσαμε δηλαδή. Κάπως πιο αρνητικά τώρα. Θεωρώ ότι παρά την ε, παρόμοια ανάλυση για το ότι είναι οξύ το πρόβλημα, για το τι προκαλεί ομοίαντο στην υγεία, Θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές ομάδες ε, δεν φαίνονται καθαρά πεπισμένες ε, ότι αν θέλουμε σήμερα να γλιτώσουμε, να σώσουμε ζωές, απαιτείται μια νομοθεσία δεσμευτική που θα πρέπει να προχωράει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και λυπάμαι, λυπάμαι που δεν πετύχαμε μια πλειοψηφία, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι τόποι ε, αποθήκευσης, αποθήκευση αμοιάντου, γιατί δεν υπάρχει ένα κατάλληλο αρχείο και κυρίως ε, ότι δεν υπάρχει, ότι θέλουν να μειώσουν ε, ε τις ε, έκθεση το όριο έκθεσης της σύνες αμοιάντου. Και θα ήθελα να σας πω και ζητάω και την στήριξή σας ε, για τις δύο τροπολογίες που με απασχολούν ιδιαίτερα, αυτή η 55 η για υποχρεωτική διάκριση ανάμεσα στον θράψιμο και στο μη θράψιμο αμίαντο, γιατί έχουμε ε, εντελώς διαφορετική επιρροή και θα πρέπει να δούμε τα διάφορα προϊόντα ε, και τα προϊόντα υποκατάστασης του αμοιάντου γιατί δεν μπορούμε να έχουμε άλλα προϊόντα που σε 5-10 χρόνια θα είναι και αυτά ιδιαίτερα βλαβερά για την υγεία. Αυτά τα δύο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ε, Ρότζερ Έλμερ και μετά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 τα ενώματα τα οποία ε, μας αναφέρεται, Υπάρχει λοιπόν αυτή η μελέτη την οποία κατέρτισαν οι εμπειρογνώμονες από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες και όλα αυτά ε, δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετρήσιμος κίνδυνος, όπως σας είπα, από τον άσπρο αμίαντο. Και νομίζω, αν θέλουν οι συνάδελφοι, μπορούν να ε, ανατρέξουν σε αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, τίθεται το θέμα, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές εκθέσεις ε, που αναφέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος, ενώ υπάρχουν και άλλες που λένε ότι δεν υπάρχουν. Ο συνάδελφός μου, ο Ντέρι Κλάρκ, αναφέρεται στην έκθεση Πίτε του 1977, όπου κάνει ένα μεγάλο σημαντικό λάθος. Αναφέρει ότι επειδή το 90% του αμοιάντου ε, είναι λευκός, ε, άρα ο καρκίνος που προέκυψε είναι από λευκό αμοιάντο. Άρα δηλαδή ε, απλά κάνει μία παραδοχή. Υπάρχουν όμως τρεις παράγοντες που μπορούν να συνδυαστούν για να αποδαιμονοποιηθεί ο λευκός αμοιάντος. Μήπως θέλετε παρακαλώ να σχολιάσετε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό είναι το θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Αυτό θα κάνω, αλλά σας εξηγώ. Ναι, αλλά κοιτάξτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ ομιλητής. Ε, εντάξει, θα συντομεύσω και ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας ε, παρέμβαση. Θέλω να πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ σχετικά με όλο αυτό το λόμπινγκ που έγινε από Αμερικανούς δικηγόρους ε, διαιτητικών δικαστηρίων. Αυτό φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Προκύπτει λοιπόν το εξής ερώτημα. Επειδή οι τροπολογίες σε μεγάλο βαθμό δεν κάνουν τη διαφοροποίηση ανάμεσα στα διάφορα είδη αμία. Μερικά από αυτά είναι τοξικά, αλλά όχι όλα. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να υποστηρίξω αυτέ τι τροπολογίε και γι' αυτό θα τι ε, καταψηφίσω. Και οποιο άλλο ε, συνάδελφο ε, συμφωνεί μαζί μου θα τον καλέσω να κάνει το ίδιο και εγώ. Ευχαριστώ. Γιώργος Μπακ και μετά ο επόμενος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, δουλειά του. Νομίζω ότι ευθύς εξ αρχής ε, προσπάθησε να συζητήσει με τους σκιώδεις συζητητές ε, και έδειξε πνεύμα συμβιβασμού. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ στην, σοβαρότητα αυτής της έκθεσης. Ε, είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας ε, και κατορθώσαμε να την προβάλλουμε και αυτό είναι καλό. Ε, εμείς καταθέσαμε ορισμένες παρατηρήσεις στις συμβαστικές προτάσεις. Αυτό έγινε από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αναφέρομαι στην καταχώρηση και στην μελέτη αντικτύπου και επίσης και στην επισήμανση σχετικά με τα προγράμματα δράσης μέχρι το 2028. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας ε, είναι ο πρωτοπόρος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την εκπαίδευση των απασχολούμενων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν προδιαγραφές, ε, υπήρξε και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμείς το επισημάναμε ιδιαίτερα αυτό. Ε, Κατά την άποψή μου λοιπόν είναι μια καλή έκθεση και λόγω της ε, καλής συνεργασίας ε, καταλήξαμε στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Κατά πρώτον να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πραγματικά ε, σκληρή προσπάθεια για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τοπολογίε και όλοι να μπορέσουν να συγκλίνουν σε κάτι. Τον ευχαριστώ πολύ λοιπόν γιατί πραγματικά το προσπάθησε πολύ. Το θέμα του αμοιάντου είναι πραγματικά σημαντικό, είναι σαφές αυτό. Και ο κυρίως εισηγητής και οι σκιώδεις καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δούμε τον αμοιόντα από την πλευρά της εργασιακής υγείας. Είμαι ικανοποιημένος λοιπόν που στο τέλος μπορέσαμε να επικεντρώσουμε το κείμενο σχεδόν εξ ε, σε, θέματα όπως οι βελτίστες πρακτικές, η εκπαίδευση, η πρόσβαση σε πληροφορίες και το καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές ώστε να εφαρμόσουν. Αυτό που πιστεύω είναι ένα εύρωστο σύνολο νομοθετικών διατάξεων. Βεβαίως, η συνολική εξάλληψη του αμοιάντου είναι κάτι που δεν με βρίσκει το σύμφωνο γιατί δεν ξέρω πώ θα υλοποιηθεί. Πάντω έγινε μια προσπάθεια να γίνει πιο ρεαλιστική η προσέγγιση μα στι ε, συμβαστικέ τροπολογίε. Είναι απαγορευμένη ουσία ο αμύαντο, προβλέπεται από την οδηγία REACH, αλλά σε λίγε περιπτώσει μπορεί να ε, ελεγχθεί εξ ολοκλήρου η χρήση του και μάλιστα για περιπτώσει όπου δεν γίνεται παραγωγή στην Ευρώπη, στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει ακόμη αμίαντος σε υπάρχοντα κτίρια, μπορεί να έχει κινδύνους για την εργασιακή υγεία, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά κινδύνου, όπως στην γεωργία. Ο αμίαντος χρησιμοποιείται σε αποθηκευτικά κτίρια, σε στέγες. Εδώ η πρόσβαση των εργαζομένων είναι σπάνια. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη. Η συνάδελφοι νομίζω με στήριξαν στα σχέδια διαχείρισης για την εξάλληψη του αμοιάντου που προβλέπονται. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι ποσοστά αμοιάντου εμπεριέχονται, πώς ε, επηρεάζει και τι είναι το καλύτερο να κάνει κανείς γιατί δεν είναι ο στόχος να ανακινήσουμε τον υπάρχοντα αμίαντο και να εκθέσουμε τους εργαζομένους σε περιτούς κινδύνους. Όμως όπου είναι επικίνδυνα τα ποσοστά περιεκτικότητα σε αμίαντο θα πρέπει να εξαλειφθούν. Δεν μπορώ να στηρίξω όλες τις συμβαστικές λοιπόν τροπολογίες των συναδέλφων που ζητούν νέα νομοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι οι φυστάμενοι είναι επαρκής στο συγκεκριμένο τομέα και θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην καλύτερη υλοποίηση και τη μεγαλύτερη στήριξη όπου χρειάζεται. Υπάρχουν και άλλα σημεία του κειμένου όμως ε, που εκεί μπορώ να στηρίξω τις ε, συμβαστικέ τοπολογίε. Όσο για τον Αμίαντο Χρυσοτήλη, νομίζω είναι πολλοί συνάδελφοι που έχουν έρθει σε σύγχυση από τις αφιλεγόμενες επιστημονικές απόψεις για το θέμα αυτό. Και το θέμα είναι ποια θέση θα λάβει κανείς στη συζήτηση για να δει κατά πόσο καταδικάζεται η ουσία αυτή ή όχι. Πάντως, υπάρχουν ε, συμβουλές επιστημονικών ομάδων να απόσχουμε καλύτερα από τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Ναι. Ε, παρακαλώ η Επιτροπή, αν τα κάνει σύντομα σύντομα θα μπορούσε να λάβει το λόγο ναι ή μήπω δεν ε, διαθέτει κάποιο σχόλιο. Κώστα Νταβίδ. Ευχαριστώ. Έχουμε κάνει τη συνεισφορά μας. Την έχετε στα χέρια σας. Δεν αλλάζει κάτι στα συμπεράσματά μας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν θέλετε να αναθεωρήσουμε το θέμα επιστημονικής πλευράς, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά θα καθυστερήσει. Η κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση είναι στα χέρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Επιχειρήσεων. Μπορούμε να τους ρωτήσουμε αν κάτι ετοιμάζεται, αν προβλέπεται αναθεώρηση της ταξινόμησης. Πέραν όμως αυτού, η νομοθεσία που έχει βασιστεί στον έλεγχο αυτών των ουσιών, των ελεγχόμενων θα έλεγα ουσιών, δεν χρειάζεται τώρα να αμφισβητηθεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Σκιώδης και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο να καθυσυχάζω την καρήμα ότι οι 55 και 97 από τις τροπολογίες της με βρίσκουν σύμφωνο. Θα συμφωνήσω με τα σχόλια του κυρίου Μπάχ και του κυρίου Μπένιν. Κρίμα που δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με την συμβαστική ΕΛ. Προσπαθήσαμε σκληρά για να καταλήξουμε σε αυτήν. Φαίνεται να μην το πετύχαμε απόλυτα το στόχο μας. Όσο για τον Αμίαντο Χρυσοτήλης. Πρόεδρε, είναι άποψη της μειονότητας ίσως και χρειάζεται παρόλα αυτά επιστημονική στήριξη αλλά υπάρχει τέτοια τοποθέτηση από τους επιστήμονες ότι είναι καρκινογόνος ε, ο λευκός αμύαντος και ότι θα πρέπει να απογορευτεί εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να υπάρχει αυτή η δυσκολία σωστή διάκριση των ειδών αμοιάντου, αλλά αυτό θα μπορούσε να λυθεί εφόσον υπάρχει καθολική απαγόρευση του αμοιάντου και η χθεσινή ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ότι ο λευκό αμοιάντος Χρυσοτήλη είναι πραγματικά επικίνδυνη ουσία. Θα παρότρινα λοιπόν του συναδέλφου να ε, δεχτούν την συνένεση ε, τη επιστημονική κοινότητα για το θέμα αυτό, για την κατάργηση όλων των μορφών αμοιάντου. Αυτά Πρόεδρε, ας δέσουμε τις ζώνες ασφαλείας μας και ας προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Πάνω σε αυτή τη βάση θα ψηφίσουμε αύριο ακριβώς και στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Τελειώσαμε με το σημείο αυτό της ημερική διάταξης. Και τώρα ο Ρουσάρτ Φάουιτ έχει το λόγο για τις 29 και τροπολογίες, την εξέτασή τους, οι οποίες και κατατέθηκαν στην έκθεσή του για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων ε, για μια ανάκαμψη, αηφορία κλπ. Είναι η πρότασή μας πρωτοβουλίας. Ήδη νομοδοτήσαμε για την έκθεση που η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εξετάζει επίσης ε, και στην έκθεση κύριο Χάουιτ. Είχαμε τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής 18 Δεκεμβρίου ημερομηνία και επίσης γνωμοδοτήσεις από την ΔΕΒ, ΦΕΤΣΕΙΝΤΑ και πολιτιστικών θεμάτων. Έκθεση που έχει να κάνει και με το θέμα της νομικής επιτροπής και γι' αυτό εφαρμόσουμε την ε, νομική οδομπέρες. Όταν έχουμε αυτά που διασταυρώνονται, είμαστε αρκετά γενναιόδοροι για τις τροπολογίες ε, που έστω φαίνεται ότι προέρχονται από αλλού και περιμένουμε την διατησία μετά την ψηφοφορία. Γιατί λένε μα ζητήθηκε να ζητήσουμε από αποδεκτές ορισμένες τροπολογίες αλλά εκφράσαμε αντίθετη άποψη στο αίτημα αυτό. Ίσως όμως θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε ορισμένες αντιφάσεις με την έκθεση του κ. Μπαλτεζάρ στη Νομική Επιτροπή πριν από την Ολομέλεια. Αλλά θα το κάνουμε έξυπνα, έξυπνα, σε συνόηση μαζί με τον εισηγητή βέβαια. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο για τις 29 τροπολογίες, τις συμβαστικές, με τις οποίες ασχοληθήκατε από τις 210 που σας είχαν ε, υποβάλει. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Ε, οι διαπραγματεύσεις ε, σε πρώτο βαθμό ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για σας, ακριβώς επειδή βρίσκονται σε, αυτό, σε αυτή τη φάση, να καταλήξετε σε μία συμφωνία με τον κύριο Μπαλτασάρη, ε, τον συνάδελφό μου στην Επιτροπή. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και θέλω να τοποδώσω τα εύσημα και είμαι σίγουρος ότι ε, θα έχουμε τελικά ένα καλύτερο κείμενο, ε, θα καταλήξουμε σε ένα καλύτερο κείμενο ακριβώς λόγω αυτού. Όπως είπατε σήμερα εστιάζουμε την προσοχή μας στις συμβαστικές προτάσεις, αλλά ε, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει το σύνολο της συζήτησης θέλω να πω το εξή. Πρώτον, έχουμε μια καλή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλουμε να τη στηρίξουμε, βεβαίως έχουμε να προσθέσουμε σχόλια, αλλά αυτό κατ' ουσίαν δεν ε, αλλάζει την κατεύθυνση που επιθυμεί να χαράξει η Κομισιόν και τη συγχαίρουμε γι' αυτό. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαφορετική θέση γιατί το φόρουμ που προσπάθησα να συστήσω στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο καταπολέμησαν οι ΜΚΟ, ήταν ένα θέμα πόλωσης αυτό. Ε, εδώ και τρία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει όμως τελικά καλή συνεργασία ανάμεσα στους άμεσα εμπλεκόμενους και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Ακούστηκαν οι απόψεις και της Κομισιόν και θεωρώ ότι τελικά βελτιώθηκε το κλίμα συνεργασίας. Θέλω λοιπόν, όπως σας είπα, να επενέσω όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ε, υπάρχει τώρα και ένας ε, νέος ορισμός, ε, ο οποίος ορισμός λέει ότι το CSR Άρα η ε, εταιρική ευθύνη, ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό το να το στηρίξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προκύψει συνένεση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι από πλευράς επιχειρήσεων ε, και ελπίζω και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανακαλύψουμε νέους ε, κοινοτικούς ενωσιακούς κανόνες αλλά να αναλάβουμε νέες ε, πρωτοβουλίες παραδείγματος χάρη οι κατευθυντήριε γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή για τις πολυεθνικές να υπάρχει καλύτερη υποστήριξη και από πλευράς επιχειρήσεων και από πλευράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπάρχει λοιπόν τεράστια υποστήριξη στο όλο το θέμα που συζητείτε και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, στηρίξει αυτήν την κατεύθυνση που μοιάζει να επικρατεί. Εμείς ε, ελπίζω αυτό να το κάνουμε και αυτή την εβδομάδα και στην Ελλομέλεια. Όσον αφορά τώρα τις συμβαστικές προτάσεις για όσους ήσαν παρόντες τη Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο θα συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε μια συμφωνία ανάμεσα στις ε, πολιτικές ομάδες που λέει ότι θα αφαιρέσουμε την αναφορά στο ε, προαιρετικό στοιχείο και στα σχετικά συνώνυμα και θα εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στο να προκύψει ε, μια ουσιαστική συνένεση στην Επιτροπή μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Με αυτό το πνεύμα ψηφίσαμε, στείλαμε το αποτέλεσμα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και οι σκιώδεις εισηγητές ε, ε, πρότειναν ακριβώς το ίδιο. Και χαίρομαι, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε 29 συμβαστικές προτάσεις. Ε, θέλω λοιπόν να καλέσω τους παρόντες να το λάβουν αυτό υπόψη τους, ότι έχουμε επιτύχει συνένεση στον τομέα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις σημαντικές προτάσεις, δεν θα αναφερθώ σε όλες, θα επιλέξω μερικές. Ο κύριος Μαν δεν είναι εδώ, αλλά θέλει διακάως να πει ότι όσον αφορά τις δωρεές από τις επιχειρήσεις, αυτό ε, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Προφανώς ε, και είναι αυτονόητο αυτό. Ε, ανησυχεί, εντάξει εγώ το έβαλα στο συμβασμό για να είναι απόλυτα ε, σαφές. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ικανοποιηθεί. Κατά τα άλλα, θέλουμε να έχουμε μια οξυδέρκεια, κυρίως στην τροπολογία ΓΑΜΑ. Εκεί ε, αξιολογούμε τις ευρωπαϊκές δράσεις, ε, καταλήγουμε ε, στο ότι ορισμένες πολιτικές ομάδες λένε αυτό θα γίνει στο μέλλον. Εν περιπτώσει όλα αυτά τα συμπεριέλευα στην συμβαστική υπαρτιμόν C. Στην D Ορισμένοι από τις συνάδελφοι θέλουν να είναι λίγο περισσότερο θετικοί ως προς τις ε, επιχειρήσεις ε, που απέφτιαν έκκληση να εφαρμοστούν στρατηγικές εταιρικής ε, κοινωνικής ευθύνης. Θέλω να σας επισημάνω ότι πράγματι μετακινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην συμβαστική ή e για το θέμα της κλιμάκωσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω, εκεί αναφέρουμε έναν κατάλογο που αφορά ε, στην ε, ε, βελτίωση προς τα πάνω. Και προβλέψαμε και τη σχετική διατύπωση για να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες. Όσον αφορά τη συμβαστική F, ένας ήθελε να αναφερθεί και το ISO του 2006. Εντάξει, εκεί κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι μια παγκόσμια προδιαγραφή ε, που αφορά την εταιρική κοινωνική ευθένη, γι' αυτό και την ε, συμπεριέλευα. Στην G, την τροπολογία εδώ πολύ σημαντικό για μας, για την Επιτροπή μας, είναι ένας κατάλογος κοινωνικών μέτρων, τα οποία μέτρα μπορούν να ληφθούν από τις επιχειρήσεις σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Επίσης, εξετάζουμε και το θέμα της έρευνας. Όσον αφορά την έρευνα νομίζω ότι πρέπει να δούμε περισσότερο το σωρευτικό αποτέλεσμα της εταιρική ε, κοινωνικής ευθύνης από το να λέμε συνέχεια και απλά ότι είναι κάτι πολύ καλό. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι άδικος ε, προς τους ε, συναδέλφους Επιτροπής Έρευνας. Την H, την τροπολογία, εκεί ασχολούμεθα με τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους οποίους επιλέγουν οι επιχειρήσεις. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία. Υπάρχει μια ομάδα που κατέληξε, αφού ερεύνησε το θέμα, έχει καθορίσει συγκεκριμένες ε, αρχές και αυτή η τροπολογία έτσι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάμε στην I, την τροπολογία I. Εκεί γίνεται αναφορά σε ε, βιώσιμα επιχειρησιακά μοντέλα. Επίσης αναφέρονται τα μειονεκτήματα. Πολλοί συνάδελφοι ήθελαν να γίνει αναφορά στα άτομα με αναπηρία αναφέρεται και αυτό στην I. Στην J, στην τροπολογία, το ΕΛΚ και κάποιοι συνάδελφοι είχαν σχέση σχετικά με το πώς θα αναφερθούμε στις υπεργολαβίες. Για μένα οι υπεργολαβίες, ε, η γενικά υπεργολαβία, αφορά κυρίως ε, την οικονομική κρίση έχει σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά συμφωνήσαμε όλοι ότι ε, το κείμενο ήταν πολύ προχωρημένο, τουλάχιστον για κάποιους ε, συναδέλφους του ΕΛΚ. Έτσι λοιπόν ε, διαγράφεται η αναφορά γενικά στην υπεργολαβία. Αυτό στην συμβαστική J, στην K, στην K, εκεί αρκετές εταιρείες ε, στη Μεγάλη Βρετανία ε, τουλάχιστον προάγουν ε, τον βιώσιμο μισθό αυτό όμω δεν μπορεί να γίνει κατανοητό σε άλλα κρατημέλη και σε άλλες πολιτικές ομάδες και γι' αυτό το διαγράψαμε το living wage για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε αυτή τη συμβαστική πρόταση. Αλλά θέλω να γραφτεί τα πρακτικά ότι εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ. Πάμε στην συμβαστική εκεί M, η L δεν υπήρχε πρόβλημα, εκεί είχα μία παράγραφο για τα συνταξιδοτικά δικαιώματα και για τον τρόπο με τον οποίο η διακοπή καταβολή συνταξιδοτικών εισφορών εκ μέρους των εκδοτών είχε αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Πώς μπορεί να ε, αρθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό αφορά βέβαια κάποια κρατημέλη, όχι όλα, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συνταξιωτικά συστήματα στα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, το αναφέρουμε αυτό στην συμβαστική N. Εκεί ενισχύουμε την υποστήριξή μας ε, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ, όπως είπα προηγουμένως. Αυτό για μένα όπως σας είπα και πριν, είναι ε, απόλυτα σαφές και είναι και το πιο συγκεκριμένο που υπάρχει. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. οι άνθρωποι του ΕΛΚ, κατ' ουσίαν και ο κύριος Μπουλάν, ε, πριν από ε, δύο ημέρες ε, είχαν διαπραγματεύσεις ε, για μια συμβαστική πρόταση και χαίρομαι που μπορώ να χρησιμοποιήσω τελικά το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του και το κείμενο που προτείνει. Πάμε στο Q, την συμβαστική Q. Ε, θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά προγράμματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα και νομίζω ότι όσοι το επιθυμούσαν θα είναι πλέον ικανοποιημένοι. Πάμε στην επόμενη, στην S. Αυτή είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής και καλούμε την Επιτροπή να καθορίσει ένα στόχο που θα προτείνουμε στους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή αντί να περιμένει ε, θα πρέπει να το προχωρήσει Πάντως ε, θα πρέπει να λάβει πιο ενεργά μέτρα, πιο σημαντικό ρόλο ε, σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι ανησυχούν ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενδεχομένω να αντικαταστήσει τι συλλογικέ ε, διαπραγματεύσει. Ο κ. Χιού κάθεται μπροστά μου, συνεργαστήκαμε και αυτό ανησυχεί όπω και άλλοι. Η τι, η επόμενη δεν έχει πρόβλημα όσον αφορά το προαιρετικό στοιχείο και τον εθελοντισμό, ε, να είναι εθελοντική η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ε, ένα τέτοιο κέντρο, άλλοι πάλι αναφέρθηκαν σε αρχές ελληνικής και όλα αυτά τα συμπεριλάβαμε στην σημαντική πρόταση D, η W. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Όσον αφορά τώρα τις ε, κρατικές προμήθειες τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ε, εγώ ήθελα να γίνει κάποια σχέση ε, μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ε, και των δημόσιων συμβάσεων. Έτσι λοιπόν τροποποιήσαμε το κείμενο για να λάβουμε υπόψη μας και τις σχετικές ανησυχίες που υπάρχουν να παραμείνει το θέμα των δημόσιων συμβάσεων μέσα στο κείμενο. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις που πρέπει να είναι βιώσιμες. Ε, το εξετάσαμε λεπτομερώς ε, και σε σχέση με την σχετική οδηγία. Αναφέρομαι στη συμβαστική Y. Εξετάσαμε το θέμα της διαφάνειας και συμφωνήσαμε ε, χωρίς κανένα πρόβλημα και αυτό εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών προδιαγραφών, ε, κυρίως του IIRC, αυτού του Διεθνούς Κέντρου Αναφοράς. Ε, εδώ γίνεται αναφορά επίσης στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην τροπολογία ΑΑ. Εκεί αν γίνεται αναφορά στον ε, διάλογο ε, και στο υπάρχον πλαίσιο τελικά καταλήξαμε σε έναν ε, συμβιβασμό. Στην συμβαστική ΒΒ εκεί εξετάζουμε το θέμα της σύγκλησης που είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την έκθεση. Πρέπει να υπάρχει σύγκληση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν ε, την ανησυχία του ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευελιξία. Και τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε τα θέματα της ε, εκπαίδευσης, η συμβαστική CC, η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να έχει σχέση με την εκπαίδευση να εφαρμόζεται στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά τη δική μου άποψη ε, μπορεί να ε, αφορά και την ε, σχολική εκπαίδευση. Πάντως πρέπει να επεκτείνεται στο σύνολο των σχολικών προγραμμάτων και χαίρομαι που καταλήξαμε σε μια συμβαστική πρόταση. Αναγκάστηκα να μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα, λέει ο μιλητής, γιατί είναι μια μακροσκελής έκθεση και έπρεπε να ληφθούν υπόψη πάρα πολλές απόψεις. Να αναφερθώ σε δύο τελικές ε, συμβαστικές. Ε, ίσως ε, πρέπει η γραμματεία να καταλήξει σε μια συμβαστική πρόταση και επιθυμώ βέβαια να αναφερθούν και πολλές απόψεις. Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικές. Το είπα ήδη αυτό στη γραμματεία. Ίσως πρέπει να βρούμε στην έκθεση σωστή θέση να ε, τοποθετήσουμε αυτές τις ε, γνώμες, αλλά η έκθεση να μην γίνει δυσανάγνωστη. Ε, ξέρω ότι η Γραμματεία θα με στηρίξει, αλλά και οι άλλες πολιτικές ομάδες, έτσι ώστε το θέμα να λυθεί το στομότερο δυνατόν. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά γίνεται σωστή αναφορά στις κατευθυντήριε γραμμές του ΟΣΑ. Και θέλω να πω στην Επιτροπή ότι επιθυμώ να διευκνήσω το θέμα μαζί τους να υπάρχουν ουσιαστικές ε, τροπολογίες, αυτές που πραγματικά αλλάζουν την ε, πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν το συζητήσω αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πριν από την καταληκτική ημερομηνία ε, να επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Η Πρόεδρος. Θα πάρει το λόγο συνάδελφος ε, για το πώς θα καλύψουμε τώρα και τις απόψεις των υπολείπων ε, επιτροπών. Έχουμε ένα, μια πρωτοκατάλογο ψηφοφορίας βάσει των τροπολογιών, ε, αλλά άλλαξαν οι συμβαστικές προτάσεις τις ε, διάφορες εκφράσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και το κατάλογο ανάλογα με το πώς έχουν εξελιχθεί αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω όλα αυτά να τα τελειώσουμε μέχρι το βράδυ, ώστε αύριο να έχουμε τον κατάλογο ψηφοφορίας. Έτσι. Αλλά και ο εισηγητής ελπίζω στη δυνατότητά του να τα κάνει αυτά. Πρώτος συνάδελφος ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι ταχυδρόμος ουσιαστικά. Και από τη στιγμή που ο σκιώδης ηγητής ο Σμπουλών επειδή είναι στο εξωτερικό δεν μπόρεσε να έλθει. Θα ήθελα εδώ να πω τα εξής εξ του ΕΛΚ βέβαια και του σκιώδης ηγητό ότι γενικά είμαστε ικανοποιημένοι για την ε, όλη προσέγγιση, για την ε, έκθεση την οποία βοήθησε ιδιαίτερα ο κ. Μπουλάν και μπορώ να πω στην Επιτροπή ότι το ΕΛΚ είναι υπέρ της συμβαστικής λύσης που προτείνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Επόμενος. Επόμενη μάλλον. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πάρα πολύ καλή δουλειά του. Αλλά επειδή όλη αυτή η εταιρική κοινωνική ευθύνη ξεκίνησε από τους, ε, ε, τις επιχειρήσεις, από τους εργοδότες, επεκτείνεται στην Ευρώπη τώρα σούσεις της κρίσης. Νομίζω λοιπόν ότι η δική μου η τροπολογία έχει σχέση με την προετοιμασία κανονισμών, κανόνων από πλευράς επιχειρήσεων ε, και με τη συμμετοχή βέβαια κοινωνικών εταίρων. Αυτό όμως δεν έγινε αποδεκτό. Ο εισηγητής θέλει ο νόμος ε, να επιβάλλει κάποιες λύσεις, να επιβάλλονται εκ του νόμου. Εγώ όμως φοβάμαι ότι ε, όταν θέλουμε να επιβάλλουμε νόμους, τότε αυτομάτως αποθαρρύνουμε όλους εκείνους που ακόμη δεν είναι πλάκησαν στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη, εφόσον πρόκειται για πρωτοβουλία των ε, εργοδοτών, αυτοί πρέπει να αισθάνονται υπεύθυνοι, αυτοί πρέπει να προετοιμάσουν την ανέβρεση λύσεων. Γι' αυτό λοιπόν λυπάμαι πάρα πολύ που δεν συμπεριλήφθηκε στη συμβαστική πρόταση αυτό το τμήμα της δικής μου πρότασης. Χαίρομαι όμως που συμπεριλάβατε στις συμβαστικές προτάσεις άλλες δικές μου προτάσεις. Ναι. Ο σκότης ε, του ΕΛΚ ε, θα μπορούσε να είχε βοηθήσει, πρέπει να το ελέγξουμε τώρα πώς οργανώνεται η όλη συζήτηση, Μπενιό και μετά ο επόμενος. Κοιτάξτε, δεν μιλάω ως ε, σκιώδη εισηγητές. Η κυρία Χίρση είναι η σκιώδη εισηγητριά μας για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω όμως ε, να αναφέρω δύο θέματα. Το ένα είναι πολύ συγκεκριμένο και το άλλο γενικής φύσεως. Το συγκεκριμένο θέμα για τις συμβαστικές προτάσεις είναι ότι δεν είμαι σίγουρος ότι ο συμβασμός δεν αφορά μόνο τις ε, προτάσεις ε, ε, ετεροδικία, αλλά με άλλα λόγια. Εγώ Πέρασα πάρα πολλά χρόνια στι ΗΠΑ και ασχολήθηκα με την ετεροδικία. Δεν θέλω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει στην ίδια κατεύθυνση. Εμεί ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με αστικές ε, υποθέσεις και διενέξει ε, με προβλήματα διαιτησία. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρχει έστω και μία αμυδρή υποψία ότι γίνεται αναφορά ε, στην ε, Α, Υπάρχει και κάτι άλλο που μοιάζει με αυτό που είπε η προλαλήσεσα, ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη ε, είναι κάτι το οποίο κατά κάποιον τρόπο το προβάλλουν επιχειρήσεις γιατί θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι κάνουν σωστά πράγματα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ ε, για πολιτικούς θεσμούς που προσπαθούν να οικειοποιηθούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα να υπάρχει μια έκθεση που να εστιάζεται περισσότερο στο να διασφαλίζει ότι οι εταιρείε εκείνες ε, οι οποίες ε, ισχυρίζονται ότι προβάλλουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη κατ' ουσίαν προβάλλουν άλλου είδους διεκδικήσεις βάσιμες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό προχωράει πάρα πολύ. Σας είπα, προσπαθούν οι επιχειρήσεις να καπελώσουν το θέμα της εταιρική ε, κοινωνικής ευθύνης ε, ε, και να παρισφρήσουν σε κανόνες που επιθυμεί να εκδώσει το κάθε κράτος οι κυβερνήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ως Σκιώδη εισηγήτρια για τους φιλελεύθερου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία. Εχθέ είχαμε μια σχετική συνάντηση και σχεδόν σε όλες τις συμβαστικέ προτάσεις μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ για αυτό το πνεύμα συνεργασία. Ο συνάδελφο Μπένιανιν έφυξε τη συμβαστική ΕΡ και νομίζω αυτή είναι η μόνη ε, πρόταση όπου εμείς έχουμε πρόβλημα. Για μας τους φιλελεύθερους είναι σημαντικό να τονίσουμε και αυτό αναφέρεται στην έκθεση πρώτον ε, η, η κοινωνική ευθύνη να είναι σε εθελοντική βάση ε, και θέλουμε να παραμείνει σε ε, εθελοντική βάση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι εδώ καταβάλλεται προσπάθεια να ενισχυθούν ε, οι όροι, οι προϋποθέσεις σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρυνθούν και άλλες επιχειρήσεις ε, να ασχοληθούν με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ε, Εάν λοιπόν υπάρχει ακριβώς αυτό το θελοντικό στοιχείο, αυτό διευκολύνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί και αυτές βρίσκουν ένα πλαίσιο ε, μέσα στο οποίο μπορούν και αυτές να ενταχθούν. Υπήρξαν αρκετές ε, τροπολογίες οι οποίες αφορούν στη συμμετοχή των εργαζομένων στην στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι αυτονόητο και έτσι και εφόσον υπάρχει ένα σχετικό πλαίσιο, είναι ευκταίο να υπάρχει συμμετοχή όλων αυτών. Υπήρξαν βέβαια κάποιες τροπολογίες όπου δεν ήταν απόλυτα σαφές ε, κατά πόσον στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, ξεχωριστός φορέας ε, που εκεί να εντάσσονται οι εργαζόμενοι που επιθυμούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Κατά τα άλλα υπήρξαν και κάποιες άλλες τροπολογίες που θίγουν θέματα που έχουν σχέση παραδείγματος χάρη με τους όρους εργασίας, ε, τους οποίους δεν τηρούν οι επιχειρήσεις. Ε, δηλαδή απλά ε, όταν οι επιχειρήσεις παραβιάζουν κάποιες ε, προϋποθέσεις. Αυτό είναι κάτι που κατά την άποψή μας δεν έχει σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αν μια εταιρεία ε, παραβιάζει τους εργασιακούς κανόνες, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε παρότι προφανώς δεν είμαστε υπέρ του να ε, παραβιάζουν οι εταιρείε τους εργασιακούς κανόνες. Εδώ όμως δεν ταιριάζει όπως σας είπα. Ελπίζω να συμφωνήσετε όλοι με τις συμβαστικές προτάσεις γιατί έτσι θα έχουμε μια νέα καλή έκθεση που θα δίνει νέα κίνητρα και θα ενθαρρύνει εκείνες τις επιχειρήσεις ε, ε, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν επιφυλακτικές θα καταλάβουν ότι εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα όλη αυτή την προσπάθεια. Η Πρόεδρος δεν ζητάει κανείς άλλος το λόγο. Ο εισηγητής και πάλι έχει το λόγο, αλλά... Μήπως η Επιτροπή θέλει να κάτι? Το Συμβούλιο μήπως? Όχι, Πρόεδρε, δεν θέλω να αποφασίσω εγώ στη θέση σας, αλλά είναι εδώ, προβλέπετε. Πρόεδρος, την Επιτροπή ή το Συμβουλίο. Την Επιτροπή. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, λοιπόν. Εάν θεωρείτε ότι έχετε κάτι χρήσιμο να μας πείτε. Και αν έχετε... Λοιπόν, Επιτροπή. Σουζαμπίρντ από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και ο συνάδελφός της. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Δύο σύντομα σχόλια για τις συμβαστικές τοπολογίες. Σε ό,τι αφορά τις φιλανθρωπικές δωρεές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση αυτές να τις καταστήσει υποχρεωτικές για τις εταιρείε. Δεν υπάρχει τίποτα στην ανακοίνωση της Επιτροπής που να υπονοεί ότι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση. Έπειτα στηρίζουμε πλήρως την ιδέα του το ISO 26.000 να χρησιμοποιείται ως μια νέα προδιαγραφή στο νέο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Το εξετάσαμε λεπτομερώς του πρότυπο αυτό όταν ε, μελετήσαμε το όλο θέμα και θεωρούμε ότι είναι εύστοχο. Κατά τρίτον, όπως ίσως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφυλακτική ως προς την ιδέα να υπάρχει ευρωπαϊκό λογότυπο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα πρέπει να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή και το διοικητικό κόστος ενός τέτοιου προγράμματος. Κάτι ε, ανάλογο προσπάθησαν να εφαρμόσουν εδώ στο Βέλγιο πριν κάποια χρόνια, αλλά δεν είχε και τεράστια επιτυχία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση από τις εταιρείε για τέτοιο σήμα, αλλά δεν θα είναι απλό ε, και θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή, θα δούμε κατά πόσον σήμερα μπορούμε να καθορίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση και με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και πάλι ο εισηγητής έχει το λόγο, κάτι όμως που με ανησυχεί, το έλεγα άλλωστε Μετά από όλη αυτή την εργασία για τις προφορικές ερωτήσεις, μια διαπραγμάτευση τώρα για τον δεσμευτικό ή όχι χαρακτήρα τους, ίσως ε, προκαλούσε ιδιαίτερη σύγχυση αύριο στην ψηφοφορία. Αν στη διαπραγμάτευση αυτή θα είχαμε τώρα μια προφορική ερώτηση που θα αντιμετώπιζε πάρα πρόβλημα εντάξει για τις συμβαστικές, αλλά να μην ε, επανερχόμαστε Διαφορετικά τα πράγματα θα μπερδευτούν ιδιαίτερα. Δεν θα ήταν καλό χειρισμό έτσι και τακτική. Γιατί θα υπάρξει ίσω ένα πρόβλημα και θα προταθεί μια προφορική τροπολογία και αν ε, αποσυρθεί, απορριφθεί, τότε θα απορρίψει το όλη τη συμβαστική λύση. Δεν είναι το σαστό και το καλό. Γι' αυτό παρακαλώ αν έχουμε συμβαστικέ προτάσει Κανονικά αναλαμβάνουμε υποχρέωση όλοι μας, ε, τουλάχιστον σε ένα τόσο κεντρικό σπουδαίο σημείο της όλης συζήτησης, για να διεξαχθεί καλά η οριστική ψηφοφορία θα πρέπει να σεβαστούμε αυτές τις ε, συμβαστικέ λύσει. Ε, μην περτάμε ακόμα περισσότερο με όλε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Έχει τον λόγο ο συνάλφο. Πραγματικά είναι δικαιολογημένη η ανησυχία σα. Και αυτό που θέλω να παρατηρήσω κι εγώ είναι ε, ότι εάν αμφισβητηθούν οι συμβαστικές τροπολογίες είναι το κατά πόσον πρέπει να συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες υποτροπολογίες ή όχι. Πάντως, σχεδόν συμφωνήσαμε με τις πολιτικές ομάδες για το ποιες τροπολογίες θεωρούν ότι πρέπει να μην συμπεριλαμβάνονται και ποιες όχι. Ευχαριστώ τον κύριο Ρή τώρα και τον που μας μετέφερε τα λόγια του κύριο Μπουλόν. Την κυρία Γιαζοβλεύσκα που ίσως δεν κατάλαβε πολύ καλά την παρατηρήση μου στην πρώτη μου παρέμβαση για την τροπολογία 47. Νομίζω ότι αν το είδατε διαγράφεται ο όρος με τη χρήση της κατάλληλης ρύθμισης. Οπότε αυτό που θέλατε επετέφθη στην τροπολογία. Δεν σας αγνοήσαμε. Ήθελα να είστε βέβαιοι ότι και να είναι σαφές. Στον κύριο Μπένιεν δεν γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι είστε δικηγόρος ή νομικός από τον τρόπο που μου τοποθετηθήκατε. Δεν ξέρω. Πάντως, στη συμβαστική τροπολογία αυτή κάναμε μια αναφορά στις τρίτες χώρες. Κάτι που ουσιαστικά άπτεται τη εδαφικότητας. Νομίζω λοιπόν ότι λίγο πολύ είπαμε αυτό που θέλατε. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε την ανησυχία σας. Και για την πατρότητα του θέματος αυτού, Θα πρέπει να το συζητήσουμε για να δούμε ακριβώς ε, τι θέλουν και εταιρείε και επιχειρήσεις. Οι ίδιοι λοιπόν οι όμιλοι των επιχειρηματιών εν μέρη ε, συμφωνούν μαζί σας και δεν σας επικρίνω που το λέτε αυτό, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει κίνδυνος να αγνοήσουμε περιοχές σύγκρουσης που μπορούν να δημιουργηθούν με άλλους τομείς πολιτικής. Δεν σας επικρίνω λοιπόν για αυτό που είπατε, απλώς ίσως να μην γνωρίζετε τόσο καλά τους ίδιους τομείς όπω εγώ. Πάντως, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που ανέφερα εγώ, βεβαίως δεν θέλουν ισχύουν ισχύουσα του τομέα αυτό να ε, καταργηθεί και να αντικατασταθεί. Αυτό που θέλουν όμως είναι δημόσια στήριξη. Θέλουν ο δημόσιος τομέας να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Νομίζω 6.000 επιχειρήσεις συμμετείχαν στην σύνοδο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και είπαν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε αυτά. Εσείς οι κυβερνήσεις δεν κάνετε περισσότερο. Κατά την άποψή μου έχουν δίκιο, αλλά ουσιαστικά το λένε. Το λένε και πρέπει να τους ακούσουμε. Υπάρχει και φοβός για την υπερβολική ρύθμιση. Και δεν λέω εγώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη, αλλά ο στόχος του κειμένου και ο δικός μου δεν είναι να κάνουμε λάθος. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Χίρς, ιδίω με την παρατήρηση για τον κοινωνικό διάλογο. Αν και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε ρητός, εφόσον περιέχεται. Λέτε, όντω, αλλά κάποιοι συναδελφοί, όπω ο κ. Μπένιν, ε, φοβούνται την υπερβολική ρύθμιση, κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις θα υπονομευτούν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι βλάπτει να το συμπεριλάβουμε, αν και συμφωνώ στην πραγματικότητα με αυτό που είπατε. Και σε ό,τι αφορά το κοινωνικό όσημα, για να απαντήσω και στον κύριο Ντόντ, να το σκεφτώ. Κύριε Ντόντ, θα έχετε παρατηρήσει, ίσως θα θέλατε να γνωρίζετε ότι και εγώ το σκέφτηκα αυτό και να πω ότι οι σοσιαλιστέ αυτό το έχουν καταστήσει απότερο στόχο του τι θέλουν να πετύχουν με την έκθεση αυτή. Δεν είναι δική μου προσωπική έκθεση σε κάθε περίπτωση, είναι έκθεση αυτή τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ πάντω μαζί σα και καλό θα ήταν να το συζητήσουμε κατά λεπτό, διότι υπάρχουν κάποιε πρακτικέ ιδέε για το πώ θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά θα ήθελε η Επιτροπή να δείξει ανοιχτό πνεύμα για το θέμα αυτό. Και τέλο, νομίζω η κυρία Χίρι το είπε πολύ σωστά. Μίλησε για ανα, αναζωγόνηση και τόνωση της όλης συζήτηση για το όλο θέμα αυτό ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δούμε ποια συγκεκριμένη ορολογία θα χρησιμοποιήσουμε. Πάντως, αυτό που συνέβη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση πριν από 18 μήνες. Αναζωογονήθηκε, τονώθηκε πάλι η συζήτηση για το θέμα αυτό πριν από 18 μήνες. Αλλά ο στόχος τώρα είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την κοινωνική εταιρική ευθύνη, να προωθηθεί προ τι επιχειρήσει και του ενδιαφερομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμμετέχουν και εκείνοι ενεργά στη συζήτηση και να αναπτυχθούν, να καλλιεργηθούν κάποιε από τι ιδέε που προέκυψαν από την ανακοίνωση. Νομίζω ότι το κάναμε αυτό και με το κείμενο μα, αυτό που επιδιώκουμε και αυτό που τελικά πετυχαίνουμε είναι να αναζωογονηθεί η όλη συζήτηση. Νομίζω απλώ να προσέξουμε στι συμβαστικέ τροπολογίε και τι σωστέ ιδέε. Αυτέ να περάσουν και α υπάρχει συλλογιστική γύρω από όλη αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι ο στόχο μα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, όντως αυτή είναι μια συζήτηση επί της ουσίας. στι 24 Ιανουαρίου λίγη τώρα η προθεσμή επιβολής τροπολογιών και η εξέταση του θέματος ε, στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο αφού ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, θα λάβει το λόγο για να παρουσιάσει τις 35 συμβασικές τροπολογίες ε, και για τους μετανάστες ε, την ε, επίδρασή τους κλπ. για τα σχετικά θέματα και είναι έκθεση πρωτοβουλίας. Έχετε τον λόγο. Zuerst einmal möchte ich Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Είχαμε 200 ε, τροπολογίες, ε, έτσι λοιπόν με τις 35 ε, συμβαστικές. Είχαμε πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω λοιπόν ότι κατορθώσαμε τελικά να έχουμε ένα πολύ καλό έγγραφο ε, το οποίο δείχνει και τι πρέπει να κάνει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως ε, σε σχέση με τους ε, μετανάστες και την αγορά εργασίας. Τώρα, όσον αφορά τις συμβαστικές προτάσεις, αναφέρονται καταρχήν ε, στην κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι ε, μετανάστες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η πρόσβασή τους στην υγεία, τα στις κοινωνικές παροχές, η πρόσβασή τους δεν είναι απρόσκοπτη. Υπάρχουν και πράγματα βέβαια που αφορούν πολύ συγκεκριμένα τις γυναίκες μετανάστριες. Επίσης ε, υπάρχουν και πολλές άλλες συμβαστικές προτάσεις που δείχνουν τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι αν θέλουμε να έχουμε πραγματική προσέλευση ποιοτικών ε, μεταναστών από τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή κοινωνία για να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί σε εμά. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ενσωμάτωσή τους σε πάρα πολλές συμβαστικές προτάσεις. Ε, καθιστούμε σαφές ότι η γλώσσα είναι ένα θέμα καθοριστικής ε, σημασίας ε, για να υπάρχει καλύτερη ενσωμάτωση. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, όπως επίσης και η πρόσβαση γενικότερα στο επάγγελμα. Και εδώ αναφέρουμε κυρίως την ανεξαρτησία, την οποία επιδιώκουν ε, πάρα πολλοί μετανάστες. Ε, πρέπει λοιπόν να στηριχθούν σε αυτή τους ε, την προσπάθεια. Υπάρχει αυτό το περίπημο, περίπημο ethical entrepreneurship, η ηθική επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προαχθεί. Επίσης, αν κάποιος ε, έρχεται από μια τρίτη χώρα σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ε, προετοιμασία δεν ξεκινάει όταν φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς ε, καλούμε και τις χώρες προέλευσης να κάνουν τα πρώτα ε, προκατρακτικά βήματα, να ενημερώσουν τους άμεσα ενδιαφερόμενες ποιες είναι οι διαδικασίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προετοιμασία λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε. Επίσης υπάρχει και μια άλλη συμβαστική πρόταση ε, που αναφέρεται εκ νέου στο θέμα της μετανάστευσης. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό ένα θέμα που σχετίζεται και με τις ε, αναταραχές ε, που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Αφρική. Είναι μια κατάσταση όπου ε, και οι δύο πλευρές ε, μπορούν να κερδίσουν ε, χωρίς ε, να χαθεί τη λύση επαφή με τη χώρα προέλευσης. Κατά τα άλλα έχουμε και ένα άλλο θέμα. Εμείς καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον είναι δυνατόν να υπάρχει ένα προαιρετικό σύστημα για τους μετανάστες. Και η ιδέα είναι ότι κυρίως ε, τα μικρά ε, κρατημέλη ε, μπορούν να προσφέρουν κάποια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Όλα αυτά προαιρετικά βέβαια. Απ' την άλλη βέβαια ξέρουμε ότι εάν κάποιος που είναι από τρίτη χώρα θέλει να ενημερωθεί σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μεταναστεύσει έχει 27 διαφορετικές προϋποθέσεις. Άρα δηλαδή ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση. Πέρα από αυτό, έχουμε και τους ε, ε, παράνομους ε, μετανάστες και αυτούς που τούνται άσυλο. Αυτοί πρέπει να βρουν θέση εργασίας λόγω της επιθυμούμενης ευκταίας ενσωμάτωσης. Και ένα άλλο θέμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ο κοινωνικός συντονισμός και εδώ λέμε ότι ε, θα πρέπει και υπάρχουν εντωμεταξύ πολλές ε, διμερείς συμβάσεις αλλά νομίζω ότι έχει νόημα ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός Αυτά με λίγα λόγια είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία έχουμε συμπεριλάβει σε συμβαστικές προτάσεις και νομίζω ότι ε, εάν τελικά ε, θεσπιστεί η έκθεσή μας, θα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση για το πώς ακριβώς μπορεί να υπάρχει μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς κυρίως στην αγορά εργασίας. Είναι φιλόδοξος ο στόχος αλλά και λογικός. Ουγγαρέντου και η κυρία στη συνέχεια. Πρόεδρε, Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Αγία για την εξαιρετική της δουλειά στην έκθεση αυτή και τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων καθ' όλη τη διάρκεια τους. Νομίζω ότι η τωρινή εκδοχή των συμβαστικών τροπολογιών πραγματικά απεικονίζει επακριβώς πώς θα πρέπει να ε, βλέπουμε τους ε, ε, μετανάστες, τους εργαζόμενους μετανάστες ε, από κοινωνικής και οικονομικής σκοπιάς. Σωστά επικεντρώνεται στο πώς θα μπορούσαν να ενσωματώνονται πιο εύκολα στις κοινωνίες οι μετανάστες εργαζόμενοι. Και αυτό φαίνεται και από την, ε, το πνεύμα ευελιξίας που επιδεικνύεται στην τροπολογία II, δύο ηλεκτρικό. Επίσης πώς θα μπορούσαν καλύτερα να ανταποκρίνονται στις ανταγωνιστικές προκλήσεις οι μετανάστες και επίσης δεν θέλω να τονίσω το πόσο επίκαιρη είναι αυτή η έκθεση. Αυτή τη στιγμή οι φόβοι για την εισαγωγή εργαζομένων ουσιαστικά ε, έχουν πυροδοτηθεί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και πυροδοτούνται, συνταυλίζονται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ πάντως για την εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών που και εμείς υποβάλαμε από το ΕΛΚ. Ευχαριστούμε η κυρία Μπλινκεβιτσούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω την κυρία Χίρς, την εισηγήτρια. Είχαμε μία σταθερή και επικοδομητική συνεργασία. Το πλέον σημαντικό είναι ότι διαρκώς αναζητούσε να επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών ομάδων. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε 35 συμβιβαστικές τροπολογίες και η δική μας ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, θα τη στηρίξει. Θα τη στηρίξει γιατί η συγγήτρια πραγματικά έδωσε μεγάλη προσοχή στις δικές μας τις προτάσεις. Εφόσον ο χρόνος πιέζει να σταθώ σε μια κεντρική ιδέα ότι στις συμβαστικές τροπολογίες προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι η καλύτερη δυνατή ένταξη γίνεται μέσω της αγοράς εργασίας. Οι μετανάστες πολλές φορές πέφτουν θύματα διακρίσεων και ως προς τις συνθήκες εργασίας τους και ως προς το μισθό τους. Επικεντρωνόμενοι στο σημείο αυτό λοιπόν, ε, ουσιαστικά ε, ε, ευχαριστούμε την προσοχή των κατωμελών στο πώς έχει η κατάσταση και λέμε ότι δεν θα πρέπει να την ε, δεχτούμε την κατάσταση αυτή. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι το τι γίνεται με τα παιδιά των ε, μεταναστών εργαζομένων. Το ερώτημα είναι, έχουν ε, τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να ενταχθούν επιτυχώς στην κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής εξ αρχής. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ και ελπίζω να τύχει στήριξη από την πλειοψηφία είναι το δικαίωμα στην εργασία. Το δικαίωμα των μελών των οικογενειών αυτών των μεταναστών να εργαστούν. Ξέρουμε ότι έχουν δικαίωμα στην απασχόληση θα έπρεπε να έχουν και αυτοί και βεβαίως αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει και από το κοινωνικό βάρος που εκπροσωπούν οι μη εργαζόμενοι. Εάν μπορούσαν να κατανεμηθούν δηλαδή, ε, εάν μπορούσαν τα μέλη της οικογένειας να αναλάβουν και εκείνοι κάποια θέση εργασία. Τώρα να θυμίσω στην κυρία Χίσο ότι το σύστημα των βαθμών των πόντων αρχικά δεν μας φαινόταν σωστό. Όμως ε, Σιγά σιγά βρήκαμε μια λύση και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει αυτά τα συστήματα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πάλι σας ευχαριστώ για την πολύ καλή σας δουλειά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω την συγκήτριά μας για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο εξέτασα την έκθεση αυτή και βεβαίως το μεγάλο αριθμό τροπολογιών που προέκυψαν. με την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και το άρθρο 50, όπου είχαμε θετικότατο αποτέλεσμα στη δική μας γνωμοδότηση, βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ καλή αλληλοσυμπλήρωση, ένας καλός αλληλοσχετισμός μεταξύ των δύο κειμένων για την καταπολέμηση της διακριτικής ε, μεταχείρισης. Αυτό νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μπορεί να στηριχθείτε. πρόκειται για ημεδαπούς είτε για αλλοδαπούς εργαζομένους. Και νομίζω ότι πετύχαμε τους συναδέλφου να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ του τι ισχύει για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι για τους πολίτες τρίτων χωρών. Ε, είναι λεπτομερέστατη η έκθεση, πιστεύω, που Κοιτάζει το τι γίνεται και στις χώρες προέλευσης, ακόμη και το τι θα μπορούσε εκεί να βελτιωθεί. Από αδίστακτες υπηρεσίες πρόσληψης, ε, επίσης η εξέταση των επαγγελματικών προσόντων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιότητες των εργαζομένων. Είναι πολλοί οι πολίτες τρίτων χωρών που δεν αξιοποιούνται είναι το αντίθετο από αυτό που είναι μάλλον το φαινόμενο της κατασπατάλησης εγκεφάλων όπως θα μπορούσαμε να το πούμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα στηρίξουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ε, ισχυρή, διεξοδική και θετική έκθεση που δεν αγνοεί τα προβλήματα ίσα ίσα να ζητά τρόπους για να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις αυτά. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν την Κάποιος άλλος, όχι. Έχετε το λόγο κύριε μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία και νομίζω ότι ε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο γιατί έχουμε ένα πολύ καλό έγγραφο που αναφέρεται ε, όχι μόνο στο παρελθόν ε, αλλά και για το μέλλον για να έχουμε μια ε, καλή νοοτροπία και στάση, μια καλή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Με το σημείο αυτό της ημερής σας διάταξης ολοκληρώσαμε την εξέτασή του και τώρα α, ναι, θα το ψηφίσουμε αύριο. Και η στο Μάρτιο τον Απρίλιο. Από την αρχή είχαμε πει ότι για το σημείο 6 η κυρία Τσίμερ δεν είπατε δεν χρειάζεται να συζητηθούν οι συμβαστικές τροπολογίες για την γνωμοδότησή της. Γι' αυτό περνάμε στο σημείο 7, 8, 9, 10, 11, 12 κοινή συζήτηση που σας προτείνουμε Πρόκειται για την απαλλαγή. Πρώτη συζήτηση για την ε, γνωμοδοτήσεις και, από, και να κάνω με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, πρώτη γνωμοδότηση, εκτέλεση γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα 3, Επιτροπή. Λοιπόν, γενική ανάλυση ξεκινώντας και χαιρόμαστε για το ότι δεν υπάρχουν λάθη και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε τις αποδόσεις των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και σχετικά με τους πολιτικούς στόχους που επιδιώκουμε και το θέμα μιας στρατηγικής μέχρι το 2020, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα πάντα. Λοιπόν, θα που το FSA με μεταφορές ανάμεσα στις γραμμές του προπολογισμού και στον διορθωτικό προπολογισμό για πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ δεν δόθηκε στους δικαιούχους το σχετικό ποσό, κάτι που περιπλέκει ιδιαίτερη τη διαδικασία και δημιουργεί κινδύνους για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Επίσης για την τεχνική αρρωγή είχαμε ένα συμπληρωματικό προπολογισμό 3,25 εκατομμύρια ευρώ, χαιρόμαστε γι' αυτό, και επίσης για την απασχόληση στο πρόγραμμα Programs. Εκεί έχουμε όμως ένα ποσό κάπως ισχνότερο, συγγνώμη ζητάει η Πρόεδρος, χαμηλότερο από τον ρόλο που κανονικά φαίνεται να παίζει και μας δημιουργεί ένα πρόβλημα αυτό. Και επίσης η εκτέλεση για τέρες είναι 74% για την ε, περίοδο 2010-2011 ενώ ήταν 67% 2011-2012. Από την Επιτροπή ζητάμε να βελτιώσει την χρήση αυτού του ποσού του κονδύλι και θα δούμε βέβαια και για ποιο λόγο θα ήθελα να αλλάξει τη βάση παρεμβαστούρες. Για τη δεύτερη τώρα γνωμοδότηση για τις ε, διάφορα ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον προπολογισμό τους, ε, τι διαπιστώνουμε ότι τα προγράμματα μέσω των Ιδρυμάτων ε, είναι προσαρμοσμένα στη σημερινή κατάσταση και στις πολιτικές προτεραιότητες και περιμένουμε να συνεργαστούν στενά αυτά τα Ιδρύματα με τις αρμόδιες επιτροπές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επεξεργασία των ετησίων προγραμμάτων τους ε, και για να είναι αποτελεσματική όλη η εργασία και ζητάμε από την Επιτροπή να κάνει όσο γίνεται καλύτερη χρήση αυτών των κονδυλίων ε, για τα ιδρύματα και για τη συνεργασία μεταξύ τους ε, και όπως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερη η λειτουργία τους ε, και η παρουσίαση των λογαριασμών από τα διάφορα ιδρύματα να γίνονται με περισσότερο μονικό τρόπο ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τις ε, αποδόσεις. Ε, τώρα το ειδικό προπολογισμό του ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, για την βελτίωση, την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης τι διαπιστώνουμε εκεί, ότι η στρατηγική μέχρι το 2020 έχει ενσωματωθεί πολύ καλύτερα και ότι το ελεκτικό συνέδριο είπε ότι οι λογαριασμοί του Σούμπης έλεγξε που ήταν σωστοί και προτείνουμε επίσης ε, να επιδοκιμάσουμε το σχέδιο για τη βελτίωση κατάρτισης για προγράμματα εργασίας και παρατηρούμε επίσης ε, για τις βελτιώσεις ε, που θα πρέπει να επιφέρουμε γιατί το 67% το 2011 Πολύ λιγότερα καταγράφηκαν όμως επισήμως στο τέλος της χρονιάς και επίσης ε, για τις πιστώσεις πληρωμών ε, λέμε ότι βελτιώθηκε η κατάσταση αλλά λυπούμεθα γιατί το ΣΕΝΤΕΦΟΠ από την άλλη μεριά δεν διαθέτει διευθυντή. Και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ διαμαρτύρεται για αυτό που λέμε αλλά γιατί όχι, δεν βρίσκω κανένα λόγο να το αλλάξουμε και να μην το συμπεριλαμβάνουμε και νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να υπαγρυπνεί καλύτερα και να παρεμβαίνει μάλιστα σε μια παρόμοια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μας. Οποιοςδήποτε κι αν είναι ο υπεύθυνο τέταρτη γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό για την κατάρτιση ETF Βλέπουμε τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου, τι λέει, ότι οι τίσχοι λογαριασμοί κηρύχθηκαν σωστοί και μετά από την ε, Αραβική Άνοιξη νομίζουμε ότι συνέβαλαν ιδιαίτερα ώστε να έχουμε ένα επαναπροσανατολισμό ακριβώς ε, της πολιτικής και της μεθόδου παρέμβασης μετά από αυτά τα μίζωνα πολιτικά θέματα και παρεμβάσεις. Εδώ επίσης ε, λόγω της απαλλαγής για την ε, υγεία και την ασφάλεια για το Ίδρυμα αυτό, στο χώρο εργασία, ε, στο θέμα αυτό, το σχετικό Ίδρυμα στην, στο Μπιλμπάο. Εδώ γιατί πρόκειται να πούμε ότι χαιρόμαθα ότι πολλά θέματα έχουν εξεταστεί για την ίδια και την ασφάλεια στον χώρο εργασία. Πρόβλημα υπάρχει μια ανάλογη κινητοποίηση της Επιτροπής σε θέματα παρόμοια και το ελεκτικό συνέδριο ότι διαπίστωσε την, το ορθόν των λογαριασμών, άρα λοιπόν χαιρόμαστε και προτείνουμε να λάβουμε υπόψη μας και την παρατήρηση του λεκτικού συνεδρίου ότι η ακύρωση από το 4% όμως πέρασε στο 8%, στο 8% το 2000, από το 2010 μέχρι το 2011 και ο προπολογισμό του Ιδρύματος για το 2011 θα είναι 0,9% ε, εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το 2010 δηλαδή. Το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την παρακολούθηση των συνθήκων ζωής και συνθήκων εργασίας, το Eurofund, Ίδρυμα του Δουβλίνου. Χαιρόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα εργασίας του Ιδρύματος του Δουβλίνου προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της κρίσης και με τις συνθήκες ε, εργασίας, όπως επίσης και με τις δυνατότητες να τονισθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ε, συγγνώμη διορθώνει η Πρόεδρος, πρώτον, τι προτείνουμε, να εκφράσουμε το υιοθέτησή μας σχετικά με τον τρόπο που υιοθετήθηκε ακριβώ ε, η προσαρμογή τους ε, για θέματα κρίσης και για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αηφόρο, αποτελεσματικό ε, δημόσιο τομέα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να δούμε και τις διαθωτικές αδυναμίες σε σχέση με αυτή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και επίσης ε, κάτι που το λεκτικό συνέδριο δεν διαπίστωσε καμία παραβίαση, αλλά να πούμε δηλαδή ότι διαπιστώθηκε ότι ήταν διάφανος ο χαρακτήρας των προσλήψεων. Αυτά και τελειώσαμε με το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Εδώ θα πρέπει να μην θεωρήσετε απλά και μόνο τυπικό, τυπική την παρουσίαση αυτή, γιατί όλα αυτά που γίνονται στον προπολογισμό έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση και αυτών των ιδρυμάτων και γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για... και στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής μας. Και sorry, και Edith μετά. Λοιπόν, πρώτα θα ήθελα σχετικά με το τμήμα 3 Επιτροπή να πω ότι συμφωνούμε με όσα υπόθηκαν από την Πρόεδρο. Θεωρούμε ότι τα διάφορα εργαλεία και η μελέτη τους είναι κάτι το πολύ σημαντικό και επίση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η πρακτική. Πολλά χρήματα παραμένουν στο τέλος. Το είχαμε τονίσει προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι το αρνητικό να μην χρησιμοποιούνται τα κονδύλια μέχρι το τέλος του χρόνου και αυτό και για το κοινωνικό ταμείο αλλά και το και τώρα βλέπουμε ότι πρόκειται για κάτι το αρνητικό εδώ. Λέμε ότι εντάξει, ναι, καλά πάνε όλα, αλλά δεν καταφέρουμε να τα δαπανίσουμε όλα αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν γιατί θέλουμε περισσότερα, μας ρωτούν. Γι' αυτό κυρία Πρόεδρε, ε, χαίρομαι που τονίσατε την πτυχή αυτή στην έκθεσή σας. Ότι τα κονδύλια που δεν διατίθενται δημιουργούν προβλήματα. Και βέβαια συμφωνώ και με τις υπόλοιπες διαπιστώσεις σας. Θεωρώ ότι υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα για τον τρόπο αντιμετώπιση ε, μερικέ φορέ των Ιδρυμάτων. Μερικές φορές αναλαμβάνονται ιδιαίτερε υποχρεώσει πολλέ υποχρεώσει για το μέλλον και σε άλλε περιπτώσει υπάρχει ένα άλλο γενικό πρόβλημα, κυρίω στα πλαίσια του ΣΕΝΤΕΦΟΠ για την όλο προγραμματισμό, ο οποίο δεν στέκεται στο ύψο του. Και η το ποιο θα πάρει τι γίνεται καμιά φορά στο τέλος, τέλος του χρόνου και αυτό ίσως σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τον σωστό ορθό προγραμματισμό γιατί εκεί παρατηρούνται διάφορες αδυναμίες και αυτό δεν είναι και τόσο θετικό επαναλαμβάνουμε. Χαίρομαι όμως το ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν, δεν παρατήρησε τίποτα το μη ορθό στην όλη διαχείριση. Αυτό είναι πολύ θετικό, δεν συμβαίνει πάντα έτσι και μπορούμε να πούμε ότι στον τομέα αυτό τουλάχιστον ε, μπορέσαμε να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Σχετικά με το Ίδρυμα του Τωρίνου και ε, επαγγελματική κατάρτισης, ε, παρακαλώ ας προσέξουμε κάτι γιατί απαντώντας ερωτήσεις η εντύπωσή μας είναι ότι η κατάσταση για τις πληρωμές των δαπανών ε, δημοσίου μας χρήσης ε, δεν γίνονται πάντα όπως πρέπει δεν συμφωνεί το Ίδρυμα του Τωρίνου και μερικές φορές ε, πρέπει να το τονίσουμε αυτό ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια συμφωνία πλαίσιο και να επιμείνουμε σε όσους έχουν σχέση με αυτό για να μπορέσουν με τη σειρά τους να ε, συνεννοηθούν, να συμφωνήσουν για τον τρόπο δαπανών. Και ακόμα για το Ίδρυμα για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασία. Αντί για το 4% ακυρώσεις υπάρχουν 8%. Καταλαβαίνω βέβαια ότι πρέπει να το σημειώσουμε, αλλά ίσως να το διατυπώσουμε καλύτερα, γιατί δεν ε, είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσει να γίνεται και στο, στο μέλλον. Εδώ όλα αυτά συνομοδοτήσεις πάντα είναι καλά, σωστά, μπορούμε να τα δεχτούμε και μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Edith Bauer και μετά Phil Bennion. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες τις απόψεις. Νομίζω ότι όλες σας οι εκθέσεις είναι ε, πολύ καλές. Θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τη λειτουργία των οργανισμών αυτών σε σχέση με τις περισσότερες από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Επιτροπής. Τώρα για την όσα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στον οργανισμό του Bilbao και ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Προσπάθησα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία να βρω διευκρινήσει και από άλλε μεταφράσεις, αλλά στις διαφορετικές γλωσσικές εκδοχές βρήκα τρεις διαφορετικές εκδοχές της διατύπωσης. Με την επόμενη μετάφραση που βρήκα κατέληξα και σε διαφορετική, σε τέταρτη. Πώς θα επιληθεί το ζήτημα αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά το ιστορικό δημιουργίας του οργανισμού αυτού. Η κατάσταση ήταν αρκετά ασαφής ως προς το ποιος θα ήταν ε, υπεύθυνο ως προς την πατρότητα του οργανισμού και το κατά πόσον θα μπορούσε να εγκατασταθεί στο Μπιλμπάο. Έχει επιληθεί η κατάσταση, έχει προχωρήσει καθόλου. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Ευχαριστούμε, Φιλμπενιό. Ευχαριστώ. Διαβάζω τις σημειώσεις της κυρίας Χάρκιν, γιατί νομίζω ότι έχει να απαντήσει στον κύριο Κάμερον, οπότε δεν μπόρεσε να παραστεί. Κατά πρώτον, ευχαριστεί την εισηγήτρια και έχει μια-δυο ερωτήσεις και κάποια σχόλια για την απαλλαγή του γενικού προπολογισμού. Ξέρουμε γιατί μειώνονται τα ποσοστά κατανάλωσης στην Eurest και κατά πόσον θα μπορούσε να αντιστραφεί αυτή η τάση, τι θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε. Ω προ το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, εκφράζει ικανοποίηση με την απόκριση του στο ελεγκτικό συνέδριο και ιδίω ω προ τα ποσοστά των αυτομάτων μεταφορών στον τίτλο 2. Τρίτον, για το Eurofound, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεω και Εργασία, ε, είναι ικανοποιημένη με τα κριτήρια που ισχύουν. Τώρα για τον όσο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, εκφράζει ικανοποίηση για την δική τους απόκριση. Βεβαίως υπήρξε κάποια σύγχυση για το κατά πόσον ήταν ε, σαφής η εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Αυτό μάλλον ε, και για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική Εκπαίδευση βρίσκει ότι είναι ικανοποιητική και η δική του απάντηση στο ελληνικό συνέδριο και τι ε, συστάσει του. Και ως προς το 2011 και το τι για αυτούς τους οργανισμούς ε, συστήνει την καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων των ε, οργανισμών αυτών στη στιγμή εκπόνησης της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων προκειμένου να αποφευθούν επικαλύψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα πριν να δώσουμε απαντήσεις όσους ε, πήραν το λόγο, μήπως υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, όχι. Τότε το λόγο έχει ο κ. Κάντος, ε, διευθυντής στην Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να πάρω το λόγο στα πλαίσια της απαλλαγής για το 2011. Εκφράζει την ικανοποίηση της ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο κεφάλαιο στη συζήτηση τη Επιτροπή σα για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αυξάνεται έτσι το ποσοστό διαφάνειας τη δημοσιονομικής διαχείρισης. Εδώ επιβεβαιώθηκαν οι δημοσιονομικές εξελίξεις των προηγούμενων ετών. Είδαμε να ε, υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες της συνολικής ε, εκτίμησης του ελεγκτικού συνεδρίου για το 2011. Πρώτα απ' όλα είναι καλύτερη η χρήση των πόρων, οι διάφορες διαδικασίες που ίσχυσαν και βεβαίως τα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόστηκαν από τα κράτη-μέλη. Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο έχει θετικότερο αντίκτυπο και κυρίως ε, ε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα δύσκολης εφαρμογής, υψηλότερου κινδύνου μάλλον. 40% του όγκου των πληρωμών αξιοποιήθηκε καλύτερα σε σχέση με το 2010. Με αυξημένη ταχύτητα. Οι συνολικές πληρωμές έφτασαν τα 10,4 δις, αν και τονίζεται στο σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής ότι 2,7 δις θα πρέπει να μεταφερθούν στις αρχές και έπρεπε μάλλον να εκταμιευθούν ε, στις αρχές του 2011 λόγω των ε, ανεπαρκών μεταφορών από το 2007-2011 ε, έχουν υποστηριχθεί από το Κοινωνικό Ταμείο 49 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες. Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν στη συνέχεια. Έτσι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχέστερα την οικονομική και κοινωνική κρίση. Θα πρέπει να είναι ισχυρό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στο μέλλον, προκειμένου να επιδιωχθούν επιτυχώς οι πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής το 2020 και στην κοινωνική πολιτική και στην απασχόληση το 19% των πόρων του Ταμείου αφιερώνοντας στις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής. Εδώ λοιπόν θα δούμε τις συστάσεις των δικών σας εκθέσεων και ελπίζουμε να συνεχιστεί η αρμονική συνεργασία μας με την Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διαθέσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, bien, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο θα προσπαθήσω να κάνω μία περίληψη της απάντησης. Κύριε δεν ε, λυπάμαι γι' αυτό. Αν δεν ήταν μέσα έτσι δεν ξέρω <laughs> πόσο καλό θα ήταν. Αλλά λέτε ότι είσαστε διαθέσή μας για να απαντήσετε. Τρία ερωτήματα δεν απαντήσατε σε κανένα ουσιαστικά κάνατε μια διαφήμιση τη Επιτροπής. Πολύ καλό αυτό, αλλά τρία ερωτήματα που τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα το θέμα της κ. Αρκίντ, δηλαδή η Επιτροπή, αυτή την εργασία των Ιδρυμάτων, μήπως σημείου τις χρησιμοποιεί για την καλύτερη εξέταση της όλης ανάπτυξης. Το ερώτημα της κυρίας Μπάουερ που έχει να κάνει με τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου και για το 15 για δύο ευρωπαϊκούς οργανισμούς που βασίζονται στην Ισπανία. Αλλά εδώ οι διαπραγματεύσει δεν ολοκληρώθηκαν. Δεν απαντήσατε τότε σε αυτό το ερώτημα. Και τρίτη ερώτηση, στην οποία ούτε σε αυτήν απαντήσατε. Η διαδικασία πρόσληψης διευθυντή για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Τρεις συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Δεν απαντήσατε ούτε σε αυτές, ούτε στην ερώτηση του κυρίου Ρή. Ίσως εν μέρη να απαντήσατε το ποσοστό κατανάλωσης των ε, χρήσεων των πιστώσεων. Να προσθέσω και μια τέταρτη, πέμπτη μάλλον, την ερώτηση για την ε, μη ορθή μετάφραση των στόχων ε, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το πώς αυτοί αντικατοπτρίζονται στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχετικό τομέα. Είναι πέντε σημεία. Είναι σημαντικά τα στοιχεία αυτά. Θα έπρεπε να απηχούνται στις ε, εκθέσεις απαλλαγής ε, της Επιτροπής ε, απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων που απευθύνονται και στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε εδώ να επιφέρουμε βελτιώσεις με τι τροπολογίες που θα υποβληθούν για τα σχέδια έκθεσης που σας έχω υποβάλει. Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου ισχύει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και να πω στο σύνολο των συναδέλφων που πήραν το λόγο ότι στο μεγαλύτερο μέρος συμμερίζομαι τις παρατηρήσει του, όπω φάνηκε και από την ανακεφαλαίωση που έκανα. Πρώτον, για την το να λαμβάνονται υπόψη τα καθήκοντα των οργανισμών στην ετήσια έκθεση επιδόσεων, έπειτα το θέμα της έδρας του οργανισμού του Μπιλμπάου, τρίτον η διαδικασία πρόσληψης ε, του διευθυντού του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, τέταρτον το θέμα της χρήσης των πιστώσεων, των πόρων του Γιούρες και έπειτα το τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γενικώ. Ελπίζω ότι δεν ξέχασα τίποτα. Όταν λοιπόν τώρα υποβάλαμε τροπολογίες ε, της 30, μάλλον όταν από τη στιγμή που ισχύει μέχρι 30 Ιανουαρίου, στι 20 Φεβρουαρίου θα δούμε στην και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού 12 Μαρτίου ψηφίζει. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό τη ημερήσιας διάταξη ε, και έχουμε τώρα το σημείο 12 Εκεί στα γρήγορα γρήγορα πριν από την συζήτηση με τον Υπουργό να σας παρουσιάσω το όλο σχέδιο με τις προφορικές ερωτήσεις τις οποίες ε, υποβάλλουμε προς ε, εξέτασή σας. Το 13-13 είναι και όχι το 12 για τις συνέπειες της πολιτικής λιτότητα για τις συνθήκες ζωής των ε, ατόμων με προβλήματα. Η αριστερά το έχει ζητήσει και εμείς ε, συμφωνήσαμε με τις αρχής διακόπτει η πρόεδρος. προφορική ερώτηση. Θα κάνω μια ανάλυση ε, ε, το πώς ε, επηρεάζουν τα πράγματα αυτές οι πολιτικές λιτότητες και η Επιτροπή με ποιο σημείο έχει λάβει υπόψη σε αυτή την κατάσταση την ειδική και επίσης να γίνει ένας έλεγχος πώς η Επιτροπή θα θέσει σε εφαρμογή την όλη στρατηγική υπέρ παρομοίων ατόμων με προβλήματα 2010-2020 για την περίοδο αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την Συμφωνία των Εθνών για τις υποχρεώσεις της απέναντι σε παρομοιά άτομα. Και έχουμε άλλο ένα ερώτημα που παραπέμπει στην εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της έκθεσης του συναδέλφου Άνταμ Κόζα που είχε να κάνει με τη στρατηγική της Επιτροπής. Έχουμε όμως το ψήφισμα το ειδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά λοιπόν Καλό θα ήταν να το αναφέρουμε αυτό για την προφορική ερώτηση. Μήπω κάποιο επιθυμεί το λόγο παρακαλώ. Μάρφη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που βάλατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Ε, συμφωνώ με αυτά που αναφέρθηκαν στην προφορική ε, ερώτηση. Νομίζω ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να ευχαριστήσουμε όλες ε, τις ε, ομάδες πίσω για θέματα αναπήρων που έβαλαν το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Σε αυτήν την Επιτροπή και γενικότερα στο Κοινοβούλιο ασχολούμεθα με τις επιπτώσεις ε, της κρίσης. Οι επιπτώσεις είναι οξύτατες, υπάρχουν πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και γενικότερα ανεργίας. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις βίαιες επιπτώσεις της πολιτικής λιτότητας στα άτομα με αναπηρία. Υπάρχει μια πολύ καλή έκθεση, σας τη συστήνω να τη διαβάσετε. Περσινή είναι του Ευρωπαϊκού ε, Κέντρου Αναπηρίας. Επιπτώσει λοιπόν σε αυτούς και η έκθεση αυτή δείχνει ότι ε, πάρα πολλοί κινδυνεύουν να... Ε, αποκτήσουν, ε, να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπτώσεις. Και αυτό εξαιτία των μαζικών περικοπών στη δημόσια δαπάνη. Και στην Ελλάδα πάνε μέχρι 20-25%, κάτι λιγότερο στην Ιρλανδία και στην Ιταλία, τις κοινωνικές υπηρεσίες όπως ε, διάφορα ιδρύματα, ε, μείον 28% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν επιθέσεις κατά του δημοσιοτομέα και δεν προσφέρονται πια υπηρεσίες ε, από κέντρα πανσχάρη αρρωγή σε κόσμο κλπ. Πολλά και διάφορα τα οποία θίγουν τα άτομα με αναπηρία και επειδή δεν ε, ανανεώνονται υπηρεσίες ε, κατοίκων πάνω χάρη και λοιπά στην Ιρλανδία υπέρ ηλικιωμένα ατόμων ή αναπήρων ε, αρκετά υψηλό ποσό στην Ιρλανδία. Από τους κύριες λόγους της κρίσης ήταν το κόστος λόγω της έλλειψης βοήθειας για μια αυτόνομη εξυπηρέτηση και άτομα που θα μπορούσαν να βοηθηθούν έτσι λόγω αυτών των αυστηρών μέτρων λιτότητος δεν υπάρχει δυνατότητες και μιλάμε και για άτομα που ε, αντιμετωπίζουν αυτά τώρα βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να στηριχθούν τα άτομα με αναπηρία και στην ε, Μεγάλη Βρετανία υπήρξε μια περίπτωση όπου επαναπροσλήφθηκε το συγκεκριμένο άτομο που είχε απολυθεί. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, πρέπει να το συζητήσουμε και εγώ απορρίπτω τη λογική που λέει ότι ξέρετε ε, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πρέπει η αθλειότητα να κατανεμηθεί σώποσα και ισόνομα. Δεν ξέρω. Ε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Δεν νομίζω ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να πληρώσουν το τίτημα. Οι πιο πλούσιοι, οι τραπεζίτες είναι εκείνοι που θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το να το συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο. Εκτός του Κοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλές ε, και σημαντικές ε, κινητοποιήσει. Ευχαριστώ. Adam Ναι, ευχαριστώ πω μερικά πράγματα σύντομα. η Επιτροπή μας θα πρέπει να το υποστηρίξει αυτό, ότι χρειάζεται υποβολή αυτής της προφορικής ερώτησης. Και χαίρομαι που η Πρόεδρος είπε ότι με όλα αυτά τα θέματα ασχολούμεθα και με την έκθεση που υθετήσαμε προσπαθήσαμε να διαχειριστήσουμε το πρόβλημα και για την Ευρωπαϊκή επίσης Επιτροπή που θεωρούμε ότι θα μπορεί να βοηθήσει τόσο πάντων περιμένοντας τα κράτη-μέλη και κάθε κέντρο να καταβάλει την προσπάθεια που πρέπει, αλλά υπάρχει μία συμφωνία του ΟΙΕ για τα δικαιώματα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εξ του ΕΛΚ προτείνω ένα νέο θέμα να προσθεθεί. Το πώς θα αφαιρεθούν τα εμπόδια για την πρόσβαση και πώς ε, η πρόσβαση ατόμων με παρόμοια προβλήματα θα μπορούσε να είναι ταχύτερη και ευκολότερη. Και ακόμα δεύτερη πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η Επιτροπή μας θα πρέπει να επιμείνει για μια πιο ορθολογική χρήση και για τα επόμενα χρόνια να έχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης για τα άτομα με αναπηρία. Και τρίτο θέμα, η έκθεση για τη σύνολο των στατιστικών. Τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, αλλά για όσους έχουν πρόβλημα αναπηρίες θα πρέπει οπωσδήποτε οι στατιστικές να είναι ακριβείς και η Επιτροπή πρότεινε τα επόμενα 7 χρόνια όλα αυτά να αποτελέσουν μία προτεραιότητα. Το ΕΛΚ υποστηρίζει 100% αυτό το θέμα σχετικά με την πρόσβαση. Ναι, για ένα λεπτό έχει το λόγο ο καθένας, γιατί ε, είναι εδώ οι υπουργοί. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα. Λάμπερ. Ε, thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι εμείς με μεγάλη μας χαρά να στηρίξουμε τις προφορικές ερωτήσεις, ορισμένα θέματα που έφυξαν τα μέλη και κάποιες οργανώσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στην έκθεση ε, πρόσβαση στη φροντίδα. Νομίζω ότι η πρόταση του ΕΛΚ είναι πολύ σημαντική με την έννοια ότι μπορούμε να έχουμε πιο υποδυτική θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτή την πολιτική, είτε πρόκειται για μεταφορά στην εργασία είτε οτιδήποτε άλλο, τότε νομίζω ότι δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Ε, όπως σας είπα λοιπόν, η δική μου η ομάδα στηρίζει ανεπιφύλακτα την ε, προφορική ερώτηση. Ευχαριστώ. Οι Ιρλανδοί Υπουργοί καταφάνουν... Α, Σάργας ναι, ναι, Γρήγορα, γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Οι σοσιαλιστές βουλευτές χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πολύ ορθή και γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα άσκημα, τα αρνητικά ή μέχρι τώρα πολιτική για παρόμοιε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά για μας αποτελεί ένα σκάνδαλο το ότι η Επιτροπή όχι μόνο δεν απαγορεύει να συμβούν παρόμοια πράγματα, γιατί στη χώρα μας, α πούμε, καταστρέφεται όλη η πολιτική η οποία ίσχυε σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Και εδώ εδώ προωθούνται μέτρα τα οποία είναι καταστροφικά πραγματικά. Γι' αυτό την προσπάθεια αυτή την υποστηρίζουμε εμείς σοσιαλιστές και ε, θα πρέπει όμως να έχουμε και ένα κάποιο ψήφισμα γιατί δεν είναι μόνο θέμα ρητορική. Ευχαριστώ. Πολύ καλά λέει η Πρόεδρος. Αυτά που συμφωνήσαμε και για τους συντονιστές για προφορική ερώτηση χωρίς ψήφισμα αυτό είχαμε πει, ίσως ορισμένες ομάδες θελήσουν να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ομάδα κοινωνικών θεμάτων. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι χωρίς ψήφισμα δεν ξέρω εκτό αν συμφωνήσουν όλοι οι συντονιστέ για κάτι το διαφορετικό, να αλλάξουν την κατάσταση μέχρι τότε. Πάντως η εντολή που μου έχει ανατεθεί εμένα είναι να έχουμε μια προθεσμία υποβολής τροπολογιών για προφορική ερώτηση. Αυτό σα είπα πιο πνεύμα κατέχει όλα αυτά και προθεσμία μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου το μεσημέρι για το κείμενο αυτό της προφορικής ερώτησης που οι διάφοροι θα μπορούσαν να παρεύουν, όπως και εγώ η ίδια ας πούμε, για το πώς θα γίνει μια φορά στις εργασίες μας και έτσι να αντιληφθούν τις εργασίες μας για την έκθεση που είχε για μας συντάξει ο συνάδελφος Κόζε. Και μετά, 21 Φεβρουαρίου, θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές και το Μάρτιο θα πάμε στην Ολομέλεια ή τον Απρίλιο και μετά το σημείο 21 της ημερήσιας διάταξης αλλά δεν είναι εδώ κύριος Το σημείο αυτό θα το εξετάσουμε στη θέση που είχε προβλεφθεί, δηλαδή το τέλος των εργασιών μας, στο τέλος της μέρας. Έχουμε το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων με τρεις ε, Ιρλανδούς υπουργού που έχουν με σχέση με μας είναι θέματα απασχόλησης, κοινωνικές υποθέσεις και όπως συνηθίζουμε θα δώσω το λόγο στον κάθε υπουργό ξεχωριστά. Παρακαλώ μην ξεπεράσουν τα 7 με 10 λεπτά το πολύ για να μπορέσουμε να υποβάλουμε και να απαντήσουν και εκείνοι και να δούμε και πώς ε, κατεχωρούνται οι αρμοδιότητες μεταξύ τους γιατί θα πρέπει να το καταλάβουμε για να προετοιμάσουν και τις ερωτήσεις τους. Ο Ρίτσαρντ Μπρούτεν, ε, Υπουργό Εργασία Επιχειρήσεων και Καινοτομιών και έχουμε τις αρμοδιότητες του και με τις ε, προτεραιότητές μας μέσω στο Αλεξάνδρου Σέρκας ε, για την κατάρτιση των ε, εργαζομένων Ρίτσαρτ Μπρίτον και μετά Τζον Μπάρτον Υπουργό Κοινωνική Προστασίας και για το να στους ασθενέστερους, του αδύναμους και ο κύριος Σιαράμ Κάνον, ε, εξωτημένος υπουργός, ε, ε, δυστυχώς ο υπουργός παιδείας δεν μπορεί να παραστεί, εκείνος τον αντικαθιστά και έχει να κάνει τώρα το θέμα αυτό με το πολιτές πλαίσιο. Είσαστε υφυπουργός σχετικά με την παιδεία, την κατάρτιση και αρμοδιότητες οτιδήποτε έχει να κάνει με την επαγγελματική κατάρτιση Άρα λοιπόν και με τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με την προσαρμογή σε θέματα παγκοσμιοποίησης. Οι κύριοι υπουργοί θα, και οι κυρίες θα έχουν το λόγο. Λοιπόν, και θα έχουμε συνάντηση στις αρχές Φεβρουαρίου και σίγουρα θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα το πρωί. Ο Ρίτσαρντ Μπρίτον έχει το λόγο. Παρακαλούμε, 7 λεπτά αν αρκετήσετε σε αυτά θα ήταν τέλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι μπορώ να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις ε, θέσεις μας. Ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχετε σημαντικότερο ρόλο να διαδραματίσετε και αυτό είναι πολύ καλό για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Επίσης ε, γνωρίζω ότι απευθύνεστε και στα Εθνικά Κοινοβούλια και τα καλείτε σε πάρα πολλές συζητήσεις που κάνετε για την απασχόληση και συναφή. Ξέρω ότι τα μέλη της Επιτροπής σας έχουν ανησυχίες ε, σχετικά ε, με τα μέτρα λιτότητας. Η δική μου κυβέρνηση ε, αναμφίβολα καλωσορίζει το σύμφωνο για την ανεργία, την καταπολέμηση ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και την ανάπτυξη. Η ε, κυβέρνησή μας ε, έχει οθετήσει αυτό το σύμφωνο και δεν αφορά μόνο την Προεδρία. Νομίζω λοιπόν η κοινή αγορά ε, κατέστησε απόλυτα σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ανταγωνιστική, έχει φέρει ωφέλη για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και πρέπει να βασιστούμε σε αυτό στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ε, η στρατηγική 2020 είναι το σχέδιο για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο προσφέρει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να συνεργαστούν για να επιτύχουν κοινού οικονομικούς στόχους και στόχους απασχόλησης Ξέρω, η Επιτροπή σα πολύ σωστά έχει υπογραμμίσει ότι τα μέτρα απασχόληση και ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνονται από κοινού, διότι αποτελούν προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη. Ε, ξέρω τη δουλειά που κάνετε ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η Ιρλανδική Προεδρία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει αυτά να ληφθούν υπόψη στις συζητήσεις. Επίσης, ε, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και το Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τις κοινωνικές αλλαγές στο πλαίσιο λοιπόν ε, του, ε, της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου προσπαθούμε να διευκρινίσουμε ορισμένα τεχνικής φύσεως θέματα του προγράμματος κοινωνικής αλλαγής και καινοτομίας ε, που προετοιμάζει τις τριμερείς συναντήσεις με το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο. Ξέρω ότι υπάρχει κάποια διαφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επ' αυτού και ελπίζω στο πνεύμα του διαλόγου να μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία. Αυτή την εποχή που βιώνουμε οικονομική κρίση και μεγάλη ανεργία σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με νομοθετικά μέτρα παράλληλα ε, προστατεύοντας την ε, βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας ε, και τη δυνατότητα της μετακίνησης των εργαζομένων που αναζητούν θέσεις εργασίας. Ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσουν στην επιδίνωση των κανόνων εργασίας. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει πει ότι επιθυμεί πρόοδο στην νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της οδηγίας που αφορά ε, στην απόσπαση εργαζομένων ε, κυρίως ε, όσον αφορά ε, την κατηγορία των ευάλωτων εργαζομένων. Ξέρω ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα που απορρέει από την πράξη ενιαίας αγοράς. Ξέρω επίσης ότι και εσείς έχετε κάνει πολλή δουλειά σε αυτούς τους τομείς και υπάρχουν δύο άρθρα τα οποία εξακολουθούν να προκαλούν πρόβλημα το 12 και το 9. Το 9 αφορά τα μέτρα ετών τα εθνικά μέτρα ελέγχου. Θα ήθελα να ενισχύσουμε, να ενθαρρύνω την Επιτροπή των των Ενετών να δημοσιεύσει την άποψή τη. Αυτό θα μπορούσε να είναι οδηγό νήμα για όλου μα. Όπω ξέρετε, ε, εμεί ε, επιθυμούμε να υπάρχει μια γενική προσέγγιση στο τέλο τη ε, Προεδρίας μα. Θέλουμε να συνεργαστούμε σε στενά με εσά, με του και ηγητέ, για να διασφαλίσουμε τη συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επί του θέματο. Η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων εργαζομένων είναι μία από τις τέσσερις ελευθερίες ε, στις οποίες βασίζεται η κοινή αγορά. Εμείς λοιπόν ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις ε, που θα στηρίζουν τους μετακινούμενους εργαζόμενους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλές φορές τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό προτείνουμε νέα νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή που θα ενισχύει την υποστήριξη και την προστασία απέναντι σε μετακινούμενους εργαζόμενους, κυρίως όσον αφορά τη διακριτική μεταχείριση. Θα καταθέσουμε νέες προτάσεις ε, και για τα δικαιώματα απασχόλησης των ναυτικών. Η ε, Προεδρία επιθυμεί πρόοδο όσον αφορά στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ε, για την πρόταση σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια για εργαζόμενους που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Επασχόληση του Κοινοβουλίου έχει ήδη εξτάσει μια σχετική πρόταση και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν μετακινηθεί πιο κοντά σε μια συμφωνημένη πρόταση. Ε, ο πρώην, η πρώην τριμερής ε, συνάντηση, η πρώτη θα γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου και θα εξετάσει αυτή την τόσο σημαντική πρόταση ε, που θα ωφελήσει, θεωρούμε, όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, προσβλέπουμε στον επάξιο ΕΝΕΣ προτάσεις από την Επιτροπή για την Προστασία των Εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Οι προτάσεις αυτή την πρόταση είναι πολύ σημαντικές γιατί θα διασφαλίσουν ότι πολλές οδηγίες ε, ε, δεν θα ε, δυσφημιστούν επειδή θα είναι τεχνικά απαρχαιωμένες με λίγη τύχη ίσως καταφέρουμε να έχουμε έτοιμη μία πρόταση σε αυτόν τον τομέα για να εξεταστεί σε τριμερή συνάντηση. Ξέρω, ε, ανησυχείτε για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ε, και την ε, οξία οικονομική ύφεση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για επιδίνωση των κανόνων. Η Ιρλανδία επίσης θα συνεχίσει να εργάζεται σε προτινόμενη οδηγία επί της αρχής ίσης μεταχείρισης ατόμων ανεξάρτητα από τις σκεπτικές πεπιθήσεις, ε, ανικανότητα, αναπηρία μάλλον, ε, φιλετική σεξουαλικές προτιμήσεις, ηλικία ε, και ε, αυτά με μεγάλη έμφαση στους ανάπηρους και στους ηλικιωμένους. Η Ιρλανδική ε, επίση θέλει να συμμετέχει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στη διαδικασία G20. χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε να υπάρχουν σχέσεις με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Η Προεδρία θα έχει διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και με τους ε, διεθνείς κοινωνικούς εταίρους ε, εν ώψη της περιφερικής συνάντησης του Διεθνούς Γραφείου ε, Εργασίας που θα λάβει τον Απρίλη στο Όσλο και επίσης να έχουμε παρουσία και στην Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας τον Ιούνιο στη Γενέβη. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Τζόαν Μπερτον, Υπουργό Κοινωνικής Προστασίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ως Υπουργός για την Κοινωνική Προστασία στην Ιρλανδία έχω έναν ευρύντατο ρόλο. Πέραν τη ευθύνη για θέματα που παραδοσιακά θα θεωρούνταν ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας και ένταξης, έχω ευθύνη και για να διαφυλάξω τα δικαιώματα των ανέργων, την πρόσβασή τους στην εργασία, την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και τις δυνατότητες ασκήσεων και μαθητιών. Μετατρέπουμε, μεταβάλλουμε το σύστημά μας στην Ιρλανδία, ώστε όσοι χρειάζονται στήριξη στο εισόδημά τους να μπορούν μέσα από άλλους δρόμους την ενεργοποίηση, την εκπαίδευση και τι μαθητείε να φτάσουν ω εκεί. Κατά την Ιρλανδική Προεδρία, λοιπόν, θα δίνω ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα αυτά μέσω του Συμβουλίου για τι Κοινωνικέ Υποθέσει. Ένα από τα σημεία στα οποία θα επιμείνει η Προεδρία είναι να συγκεντρωθούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων το Φεβρουάριο για μια άτυπη υπουργική συνάντηση. Το γενικό θέμα θα είναι στήριξη των ε, ανέργων προκειμένου να φτάσουν στην απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία των νέων και το θέμα της εγγύησης, του Ταμείου Εγγύησης για τους νέους. Ελπίζω ότι και η Πρόεδρος και αρκετοί βουλευτές από την Επιτροπή, μάλλον γνωρίζω ότι οι Πρόεδρος και πολλοί βουλευτές από την Επιτροπή σας έχουν κάνει σημαντικό έργο για το θέμα αυτό. Η όλη συζήτηση για την εγγύηση για τους νέους ε, στην άτυπη συνάντηση θα συμπληρώσει τις επίσημες συζητήσει τη Βρυξέλλες και ελπίζουμε να υπάρξει έγκριση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πρέπει να πω ότι η πρόεδρο ε, κυρία Μπερές, έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να έρθει στην άτυπη υπουργική συνάντηση του Δουκλίνου. Επίσης θα συζητήσουμε για τις υπηρεσίες δημόσιας απασχόλησης στην Ευρώπη, για τις δεξιότητες, τα νοικοκυριά όπου πλήττονται από την ανεργία, την ε, ένταξη των ε, γυναικών μεγάλης ηλικίας στην στο εργατικό δυναμικό και την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στην κοινωνική πλατφόρμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, ω προ την εγγύηση για του νέου, έχω ορίσει το θέμα αυτό ω μια από τι προτεραιότητέ μου, διότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποκριθεί στην απειλή τη υψηλή ανεργία, που πλήττει ιδίω του νέου και σήμερα αλλά και στο μέλλον. Θα συμβεί. Είναι μεγάλες επιλογές από την ανεργία των νέων και θα μείνουν μαζί μας για δεκαετίες εάν δεν αντιδράσουμε άμεσα. Τα στοιχεία ανεργίας για την Ευρωζώνη και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά δείχνουν μια ζωφερή εικόνα, ιδίως όσον αφορά τις χαμηλότερες ηλικίες. Θέλουμε να φτάσουμε σε συμφωνία για το κείμενο όσο το δυνατόν πιο σύντομα, προκειμένου να συμβεί αυτό και να υπάρξει συμβιβασμό. Αναγνωρίζουμε ότι διαφορετικέ απόψει θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τι διαφορετικά σημεία αφετηρία του κάθε κράτου μέλου. Η πολυμορφία των θεσμικών συστημάτων και η δυνατότητα των ε, συμμετεχόντων ε, στην αγορά εργασία μαζί με τι περικοπέ και τι πιέσει σε δημοσιονομικό επίπεδο και επίπεδο προπολογισμών πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα χρειαστούν δράσει και δεσμεύσει από τα κράτη-μέλη ώστε να υλοποιηθεί το Ταμείο και η εγγύηση δηλαδή και να υπάρξουν σύντομα χειροπιαστά αποτελέσματα. Πραγματικά καλωσορίζουμε εδώ το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και την αφοσίωση που έχει δείξει στην εξετασή του, καθώ υπήρξαν πολλά ψηφίσματα τα τελευταία χρόνια και ακόμη πιο πρόσφατα στη συζήτησή σα στο Στρασβούργο την περασμένη Δευτέρα το βράδυ. Το Κοινοβούλιο θα έχει σημειώσει την πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου που να μην είναι δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Στόχος της προεδρίας μας παρόλα αυτά είναι να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη-μέλη ταυτίζονται με τους στόχους και τις πολιτικές που προτείνονται στο κείμενο για την ανεργία των νέων και ότι θα υλοποιήσουν όλα αυτά προς όφελος του πληθυσμού της νεολαίας. Πραγματικά αναμένουμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου για την εγγύηση για τους νέους και θα ληφθούν αυτές οι υπόψεις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν περατώσει το Συμβούλιο το κείμενο της σύστασης. Τώρα, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους πλέον μειονεκτούντες, Όπω θα γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει πρόταση για ένα νέο σύστημα βοήθειας για τους πλέον μενακτούντες πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει σκοπό να φτάσει σε συμφωνία στο Συμβούλιο και βεβαίω με τη συμφωνία του Κοινοβουλίου να επιτρέψει την υλοποίηση αυτού του κανονισμού μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014. Το επίπεδο τη χρηματοδότηση είναι προφανώ ε, κάτι που εξαρτάται από το επιτυχημένο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ούτω ή άλλω. Παρ' όλα αυτά, αυτό θα, το πρόγραμμα θα διαδεχτεί το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστημιστική βοήθεια. Η νέα πρόταση δεν θα καλύπτει μόνο, μόνο την επιστημιστική βοήθεια, εμπεριέχει μια απέτηση οι φορεί να προσφέρουν στήριξη για συνολικότερη κοινωνική ενσωμάτωση. Η Προεδρία δεσμεύεται να συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στι διαπραγματεύσει προκειμένου να καταλήξουμε σε μια απόφαση όσο το δυνατόν συντομότερα. Όλα τα συστήματα κοινωνική προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται πιέσει από την γύρανση του πληθυσμού. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί ή προβλέπονται από τα περισσότερα κράτη-μέλη σκοπό έχουν να στηρίξουν τα συμπληρωματικά συστήματα. Γι' αυτό κατεπήγει να βεβαιωθούμε ότι οι κανόνε που διέπουν τη λειτουργία των συστήματων αυτών υποστηρίζουν την κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών. Η προτινόμενη οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσει για την στήριξη της κοινοτικότητας των εργαζομένων με την θεμελίωση και την διαφύλαξη συμπληρωματικών συνταξιδοτικών δικαιωμάτων, η λεγόμενη οδηγία μεταφοράς δικαιωμάτων. Είναι κάτι που συζητείται εδώ και κάποια χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμη υπάρξει συμφωνία. Εμεί θα επιτελέσουμε σοβαρέ προσπάθειε ώστε να, επιτευχθεί πρόοδο διότι πραγματικά γίνεται κατεπίγουσα η ανάγκη για μια τέτοια οδηγία. Η κινητικότητα στην αγορά εργασία είναι κάτι που γίνεται όλο και σημαντικότερο λόγω τη οικονομική κρίση, των υψηλών επιπέδων ανεργία και των ανισοτήτων στι ευκαιρίε πρόσληψη ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, τα συμπληρωματικά ε, συνταξιδοτικά δικαιώματα γίνονται όλο και πιο σημαντικά και σε, ε, σε αριθμητικό επίπεδο, αλλά και σε ε, σχετικού όρου σε πολλά μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επηρεάζουν πραγματικά την κινητικότητα των εργαζομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψήφισμα τον Ιανουάριο του 2011, το γνωρίζω, αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν για να βεβαιωθούν για τη δυνατότητα μεταφορά των συνταξιωτικών δικαιωμάτων. Το να βασιστούμε στο έργο τη Κυπριακή Προεδρία είναι κάτι για το οποίο είμαστε αποφασισμένοι, καθώ και να προωθήσουμε το ντοσιά αυτό με εντατικέ συζητήσει σε επίπεδο των αρμόδιων ομάδων εργασία του Συμβουλίου. Όπω είπε ο συνάδελφό μου, ο Υπουργό Μπρούτον, η Ιρλανδική Προεδρία θα επιδιώξει το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων να διδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία του εξαμήνου. Θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι πραγματικά σφαιρική η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλου του συμμετέχοντε ότι ένα ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για το εξάμεινο είχε ήδη υποβληθεί πριν το τέλο του 2012. Τώρα, ο χάρτη τη Ιρλανδική Προεδρία για το εξάμεινο τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ε, παρακολούθηση αναχώρα, καθώ και την ανάγκη να αναλάβουν εδώ τι ευθύνε του στα κάτι μέλη για τι διαδικασίε επιτήρησης. Τώρα για το πακέτο, τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις. Ξέρω ότι δεν θα πρέπει η οικονομική κρίση που μας πλήττει να μας ε, ε, παρασύρει ε, την προσοχή και να μας κάνει να ξεχάσουμε την κοινωνική διάσταση. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με του τραπεζίτε και τι τράπεζε. Δεν αφορά αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά του πολίτε. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχέδια να προβλέψει μια δέσμη μέτρων για την κοινωνική ένταξη το Φεβρουάριο το Φεβρουάριο προτιμάνω να συμπληρώσει το ε, πακέτο για την απασχόληση της περασμένης χρονιάς. Θα δούμε συγκεκριμένε πτυχέ τη δέσμη αυτή μέτρων, ώστε να είναι μια σοβαρή δήλωση ότι η κοινωνική πολιτική είναι εξίσου σημαντική και αναπόσπαστο κομμάτι τη Ευρώπη του 2020, προκειμένου η Προεδρία να αποκριθεί στι νέε ανάγκε. Και νομίζω ότι θα απεικονίσουμε και τι δικέ σα προτεραιότητε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και εσά, κυρία μου, και του συναδέλφου. Ευχαριστούμε τρίτος υπουργός, Σχεραν Κάνων, υφυπουργός, υπεύθυνος για την εκπαίδευση και παιδεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, με χαρά να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ατλαντικής Προεδρίας για το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και τα δύο αυτά ζητήματα έχουν να κάνουν με τα επιτεύγματα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουν καθοριστεί σε στρατηγική της για το 2020. Και βεβαίως για το θέμα της Ατλαντικής Προεδρίας που είναι σταθερότητα, οι δουλειέ και η ανάπτυξη. Η συμφωνία για τις τεχνικούς κανονισμούς σε τομεακό επίπεδο, αλλά και για τον προπολογισμό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι καθοριστική σημασία προκειμένου να έχουμε την ζωτική χρηματοδότηση που θα πρέπει να διατεθεί ω το 2020 προκειμένου να επιδιώξουμε του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δύο αυτά ταμεία είναι καθοριστικά εργαλεία για την επιδίωξη ευρωπαϊκών στρατηγικών όπω νέε δεξιότητε για νέε δουλειέ, ε, η νεολαία σε κίνηση και η πρωτοβουλία για τι ευκαιρίε για του νέου. Συμπεριλαμβανομένη για του νέου. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να τονίσω ότι το Ταμείο αυτό συζητιέται στο Συμβούλιο ως μέρος του συνολικού πακέτου για την πολιτική συνοχή. Υπάρχει μια ε, μερική και γενική προσέγγιση που έχει επιδιωχθεί στο Συμβούλιο για μέρη των ε, κανονισμών συνοχής συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Ταμείου. Η συνάδελφός μου, ε, ο συνάδελφος μου μάλλον, υπεύθυνο υπουργό για τα δημοσιονομικά και τι μεταρρυθμίσει, σήμερα παρουσιάζει το Ταμείο για τη Συνοχή στην Επιτροπή Ρέντιο του Κοινοβουλίου. Η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου έχει επιτρέψει να προχωρήσουμε στι συζητήσει για του κανονισμού περί συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Ταμείου. Και έτσι μπόρεσε να ξεκινήσει τι συζητήσει το, το Συμβουλίο με το Κοινοβούλιο σε επίπεδο τριμερού διαλόγου και για τι δικέ του μέρημνε σε σχέση με το Κοινωνικό Ταμείο. Ήθελα λοιπόν να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για το πνεύμα συνεργασία που έδειξαν στι διαπραγματεύσει για τον κανονισμό αυτό ω σήμερα και για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην ε, ε, συγκέντρωση προγραμμάτων και θεμάτων όπως και αυτά έχουν συζητηθεί ως σήμερα. Κάποια από τα σημαντικότερα σημεία αφορούν το πεδίο που καλύπτει το Κοινωνικό Ταμείο και τις προτεραιότητες επενδύσεων στις οποίες θα αφοσιωθεί το Κοινωνικό Ταμείο στην περίοδο 2014-2020. Αναζητώνται ε, συμβαστικές λύσεις σε βασικά ζητήματα και είναι βεβαίως μια μεγάλη πρόκληση αυτή, αλλά είμαι πεπισμένο ότι υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω πρόοδο κατά την Ιρλανδική Προεδρία. Ενώ κάποια σημαντικά ζητήματα απασχολούν το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακόμη, σας διαβεβαιώ όλους στο Κοινοβούλιο ότι θα σεβαστούμε τη συνήθι νομοθετική διαδικασία. Τώρα για το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, να τονίσω ότι το μέλλον του Ταμείου αυτού έχει να κάνει με το τι αποφάσει θα ληφθούν τελικά και στην ενεργή διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τονίζω ότι το Ταμείο αυτό προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση ακόμη βρίσκεται επιτάπητο. Το Συμβούλιο εξετάζει το όλο θέμα εδώ και ένα χρόνο. Συγκεκριμένε προτάσει για συμβαστικέ λύσει υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια τη Κυπριακή Προεδρία απηχώντα όλε τι ε, προτεραιότητε του Κοινοβουλίου, τι οποίε ημερίζεται και εν μέρη εξετάζει το Συμβούλιο. Κάποιε από τι μέρημνε αυτέ αφορούν το πεδίο που θα καλύπτει το Ταμείο Προσαρμογή, καθώ και το τι κατηγορίε εργαζομένων θα μπορούσαν να ωφελούνται από ένα τέτοιο μελλοντικό ταμείο. Ε, έχουμε δει την έκθεση τη Επιτροπή σα για το ταμείο αυτό και πραγματικά αναμένουμε με αισιοδοξία την πρόοδο που θέλουμε να επιτελέσουμε κατά τη διάρκεια τη προεσδία μα όλα αυτά τα θέματα. Είμαστε πεπισμένοι ότι το τοπίο για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θα γίνει σαφέστερο κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν ληφθούν αποφάσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε στο Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για ζητήματα που εκκρεμούν. Προκειμένου και το Συμβούλιο να ξεκινήσει να συζητά μαζί μα τη διαδικασία τη προώθηση προς μια οριστική συμφωνία του φακέλου αυτού. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλου σα για τι ε, σαφεί παρουσιάσει σα. Και τώρα το λόγο έχουν οι δύο συντονιστέ που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσει και μετά οι υπόλοιποι. Τσαβαωρή και ο επόμενος. Από το ΕΛΚ ο πρώτος λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες που μας ήλθαν από την Ιρλανδική Προεδρία. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα τις προτεραιότητες που διατυπώσατε πριν από λίγο και να σας πω ότι θεωρούμε εμείς οι ίδιοι ότι έφτασε η στιγμή, είναι η κατάλληλη στιγμή να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με θέματα λιτότητας και ανάπτυξης. Πρόκειται για μείζον πρόβλημα σε όλες τις Ευρωπαϊκές Ένωσης και εδώ επίσης την Επιτροπή μας πέρα από πολιτικές ομάδες θα σας εγγυηθούμε ότι θα τύχετε ιδιαίτερη στήριξη ε, και για τη στρατηγική του 2020 και για την απασχόληση που αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Επίσης ακούσαμε να μιλάνε για την κινητικότητα και αυτό είναι σημαντικό. Η κυρία Υπουργό μίλησε επίσης για το θέμα της κινητικότητας. Ε, αλλά παρακαλώ προσέξτε, υπέρχει άλλη μια διάσταση στη συζήτηση αυτή μετά από την οδηγία Θεωρούμε ότι η κινητικότητα και η προστασία όμως δεν είναι πάντα κάτι το σαφές και ισορροπημένο. Και υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις στο θέμα αυτό. Χαιρόμαθε χαιρόμεθα που ανάμεσα στα σημεία της ημερήσιας διάταξης εσείς καλύψατε το σύνολό τους όλων αυτών που είναι σημαντικά. Πάντως να προσέξουμε κάτι να προσέξουμε ένα πρόβλημα που προέκυψε. Είναι ένα θέμα μάλλον τεχνικό. Είναι η δημογραφική στατιστική. Και είχαμε μια πρόταση από πλευρά της Επιτροπής Ευρωπαϊκής, η οποία όμως δεν θέλει να δεχτώ στις ε, βασικές συνθήκες ε, όλα αυτά θα έχουν ε, θα επηρεάσουν την κατάσταση και για τις λήψεις αποφάσεων και για την κατανομή αρμοδιοτήτων εδώ. Πάντως να το προσέξουμε γιατί αποτελεί σίγουρα ένα πρόβλημα και θα πρέπει να δούμε για μια ικανοποιητική απάντηση από επαγγελμής πλευρά, η οποία όμως θα έχει σημαντικές πολιτικές επιρροές. Ακούστε, θα μπορούσαμε αυτό το πρόβλημα να το εξετάσουμε και να σας το εκθέσουμε καλύτερα, να το δείσουμε περισσότερο και όχι πέρα από αυτή τη στιγμή. Κάτι ακόμα σύντομο. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Λοιπόν, κύριε Υπουργός, θεωρούμε ότι η όλη εγγύηση Ναι, αλλά πάνω από δύο λεπτά μιλάτε. Όχι ο ίδιο να πάρετε και άλλα, τόσα επτά λεπτά όσα πήραν και οι υπουργοί. Άντε, ένα λεπτό ακόμα λοιπόν. Λοιπόν, η ολιγγύηση όπως είπαμε είναι σημαντική και το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να προσέξουμε τη διαφάνεια και ακόμη κάτι για την επισητιστική βοήθεια. Θα αναφερθούμε σε αυτή σήμερα το απόγευμα. Θεωρούμε πίσω ότι είναι κάτι το σημαντικό και καλό θα ήταν εάν τα θέματα αυτά από τα, ε, και δεν μειωνόταν η σημασία των ε, κονδύλιων. Ε, για τα υπόλοιπα νομίζω τα καλύψουν οι συναδελφοί. Εντάξει. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Σάρκας για, Σάρκας για δύο λεπτά, έτσι, για να μην καθυστερήσουμε, σας παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε οι δύο κύριοι και η κυρία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία εξ ονόματος των ε, Ισπανών Σοσιαλιστών και να σας πω ότι ελπίζουμε ιδιαίτερα το 2013 να αποτελέσει πραγματική αλλαγή γιατί μέχρι τώρα τα πράγματα είναι καταστροφικά στην απασχόληση σε κοινωνικά θέματα και δεν υπάρχουν και λύσεις, έτσι κ. Μπρούτον ε, μίλησε για την στρατηγική 2020. Πεπισμένοι είμαστε ότι αν αυτή η πολιτική λιτότητα δεν αλλάξει με μόνο ε, λιτότητα και δεν έχουμε και πάλι τις ιδιαίτερες επιδιώξεις τις παλιές να είναι κάτι το σημαντικό η Ευρώπη ποιοτικά κλπ. Διαφορετικά δεν θα έχουμε ούτε προς την κοινωνική προστασία ούτε απασχόληση τίποτα. Διαφορετικά λοιπόν ε, μεγάλη καταστροφή. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει πλέον και θα πρέπει, δεν, ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες και άλλες προεδρίες ε, να συνεχίζεται αυτή η ανισορροπία γιατί από ε, μακροοικονομικής ε, προοπτικής να ελπίσουν ότι μια στιγμή αργότερα θα φτάσει η επασχόληση Όχι, θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα σε εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις ε, συμβουλευτικών. Και να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα υποστηρίξετε τη νέα στρατηγική υγείας και ασφάλειας στο χώρο η οποία ολοκληρώνεται φέτος και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα ακολουθήσει η νέα πολιτική γιατί αυτή τη στιγμή μόνο περικοπές, περικοπές, τίποτα άλλο και ξεχνάει κανείς τον κόσμο που επηρεάζεται από όλα αυτά. Θα υπάρξει μια στρατηγική και η κυρία Υπουργό τι θα γίνει, θα κάνει το Φεβρουάριο και να ακούσει και τα αιτήματά μας για τα 30 χρόνια που να ισχύουν για όλους και εδώ στο Κοινοβούλιο. Τα κράτη-μέλη ε, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα πάνω σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Τρίτος, Τζόρντε Μπαχ και μετά θα απαντήσουν οι κύριοι Υπουργοί. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε τρία θέματα. Καταρχήν στο φιλόδοξο πρόγραμμα της Ιρλανδικής Προεδρίας, το οποίο και χαιρετίζω. Νομίζω ότι ε, με τα βασικά θέματα που προβάλλατε, πράγματι θέσατε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Υπάρχει κάτι που ίσως ε, να μην σας αφορά άμεσα, αλλά το έθιξε ο κύριος Υφυπουργό. Πρόκειται για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά την άποψή μου πρέπει ως Ιρλανδική Προεδρία να αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό και κατά τα επόμενα έτη οφείλουμε να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια έτσι ώστε να ασκήσουμε κυρίως ε, κοινωνική πολιτική. Γιατί για μένα είναι λάθος ο κόσμος. Ε, κάτι δεν πάει καλά το να ε, πρώτα γίνεται εξοικονόμηση κονδυλίων και μετά να καθορίζονται οι στρατηγικές όπως η στρατηγική 2020. Κατά τη δική μου άποψη τα κονδύλια πρέπει να ταυτίζονται με τις πολιτικές που επιδιώκουμε. Το δεύτερο είναι ότι χαιρετίζω αυτό που είπατε, ότι η κρίση δεν μπορεί να αποτελεί πρόφαση για θέματα υγείας και ασφάλεια ε, στη θέση εργασία. Ε, καλό αυτό που θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί ε, θα ψηφίσουμε για την έκθεση Αμιάντου, σημαντική έκθεση αυτή και εκφράζονται πολλά αιτήματα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Τρίτο θέμα, εγγύηση για τους νέους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην ανεργία των νέων. Η ανεργία γενικότερα αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζω λοιπόν ότι στον τομέα των εγγυήσεων θα επιμείνετε, διότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν επιθυμούν να δεσμευτούν. Δεν επιθυμούν ούτε καν να ακούνε τη λέξη εγγύηση. Αν όμως εμείς ε, δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε απλά ε, θα περιοριστούμε σε κενά λόγια θα αναλαμβάνονται ίσως κάποιες ε, πρωτοβουλίες από μεμονωμένα κρατημέλη, αλλά με καμία εγγύηση. Ελπίζω στον τομέα αυτό να σημειώσετε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Εντάξει για δύο λεπτά και μετά Υπουργή. Χίρς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε και εκ μέρους των φιλελευθέρων ε, το ότι ήρθατε σήμερα εδώ. Δείξατε πολλά θέματα. Ε, υπάρχουν βέβαια πολλά θέματα σημαντικά μπροστά μας. Εγώ παρόλα αυτά θέλω να θίξω κάποια στοιχεία. Εμείς ως φιλελεύθεροι θέλω να σας πω ότι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα αναδιάρθρωσης και τα μέτρα λιτότητας. Τα θεωρούμε απαραίτητα για να επανέλθει η ανταγωνιστικότητα σε κάποια <clears throat> Παρόλα αυτά βέβαια οφείλουμε να μεριμνήσουμε στο να υπάρχει κάποια ισορροπία και να δοθούν και κίνητρα ανάπτυξης. Και από την άλλη βέβαια Θεωρούμε ότι η θέση εργασίας είναι κάτι που αφορά όλους. Πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον οι ίδιες οι επιχειρήσεις δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οι επιχειρήσεις είναι εκείνες ε, που δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης και εμείς ως πολιτικοί απλά καθορίζουμε το πλαίσιο. Σωστό και αυτό που είπε ο συνάδελφος κύριος Μπαχ, η ανεργία δεν αφορά μόνο τους νέους, όμως ε, για μας είναι πολύ σημαντική αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το, εξο... το εξής. Αν ένας νέος ε, δεν έχει εργαστεί ποτέ, τότε ε, και κατά επόμενα έτη θα είναι πολύ δύσκολο για τον λόγω του βιογραφικού του, να βρει θέση εργασίας. Οι νέοι λοιπόν, οι οποίοι δεν εργάζονται τώρα, δύσκολα θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ε, και στην απασχόληση. Αυτό το πρόβλημα θα μας απασχολήσει κατά επόμενα 20-30 έτη, άρα για μας, για τους φιλελεύθερους, είναι θέμα προτεραιότητας. Και γενικότερα η απασχόληση αλλά και το πλαίσιο για να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας. Ευχαριστούμε. Ο κάθε υπουργό από τρία λεπτά παρακαλώ. θέμα για την εξέταση της ανάκαμψης της και γενικότερα ακόμα για την ε, κυρία Μπάρτομ για τα διάφορα δικαιώματα και για την ασφάλεια και για το ε, Από αυτά θα ήθελα να ακούσουν μια κάποια πρωτοβουλία από πλευρά Συμβουλίου. Η παριστάμενοι, κύριο Σωρή, ρώτησα κάτι σχετικά με τη δημογραφική στατιστική. Καταλαβαίνω δεν είναι κανείς αρμόδιος από εσά ε, για τις στατιστικές. Μήπως λοιπόν θα μπορούσε να υποβληθεί το ερώτημα σε άλλον αρμόδιο υπουργό. Έχετε το λόγο. Μπρίτον για τρία λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω από όλες τις παρεμβάσεις φάνηκε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από μια απλή δημοσιονομική σταθερότητα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες για την απασχόληση και αυτό φάνηκε και από τις προτεραιότητες του διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είμαστε πολύ ελαστικοί και από την πλευρά τη Προεδρία, γιατί στη χώρα μα έχουμε αναγνωρίσει την ε, ανάγκη να προσαρμοστούν οι τραπεζέ μα ώστε να υπάρξουν εμπορικέ ευκαιρίε σε επίπεδο επιχειρήσεων. Μια μικρή ε, οικονομία να αρχίσει πάλι να εμπορεύεται. Χρειάζονται τέτοιου είδου παρεμβάσει. Βεβαίω ε, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εδώ θα πρέπει να προωθήσουμε για να υπάρξει ανάκαμψη. Αλλά είναι μεγάλη πρόκληση αυτή την περίοδο και θα πρέπει να εξισορροπήσουμε κάπως το πώς τοποθετούνται το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ και το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Προφανώς. Είναι μεγάλη σημαντική, είναι μεγάλη προτεραιότητα η ασφάλεια της εργασίας και του συστήματος υγείας ταυτόχρονα ένα τέτοιο εύρωστο περιβάλλον μαζί με, καλό, με καλές εργασιακές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές για την ανταγωνιστικότητά μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι όταν πιέζεται η ανταγωνιστικότητα τέτοιου είδους αρχές θα πρέπει να υπονομεύονται ή να υποβαθμίζονται. Θα σημειώσω τις διαφορές που αναφέρατε. Όντως, σε σχέση με τις δημογραφικές στατιστικές υπάρχουν αποκλήσεις. Σημειώνω σε από κύριο Σωρή. Δύσκολα εδώ θα αποφύγουμε τις διαφορές απόψεων, όμως ως Προεδρία θα αναζητήσουμε και ένα κοινό έδαφος συνεννόησης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπέρτον. Σε ό,τι αφορά την αναφορά του κυρίου Ωρη για την κοινοτικότητα των εργαζομένων και την ανάγκη να έχουμε μεγαλύτερε επιτυχίες στον τομέα της μεταφοράς των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Εδώ βλέπουμε ότι μεγαλύτερος αριθμός πολιτών των κρατών μελών ζουν ένα μέρο τη ζωή του, εργαζόμενοι σε άλλο κρατό μέλο. Και κάποιε φορέ μπορεί και να επιστρέψουν στο τέλο στην ε, χώρα καταγωγής τους. Είναι σημαντικά τα συμπληρωματικά συνταξιδοτικά δικαιώματα, προκειμένου να έχουν μια ικανοποιητική σύνταξη οι πολίτες. Είναι δύσκολο το θέμα, αλλά επιδιώκουμε να επιτελεστεί πρόοδο και εδώ. Σε όσα είπε ο κύριος Σέρκας για τις ανισότητες. Νομίζω αναφερθήκατε στις μαθηματικές εξισώσεις της οικονομίας. Όντως, το έλλειμμα στην ζήτηση είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Αλλά εδώ μιλάμε ε, για θέματα κοινωνικών υποθέσεων σε μια αρμόδια επιτροπή και είμαστε και τέτοιοι υπουργοί στην Ιρλανδία. Ο ρόλο τη κοινωνική προστασία, αν θα μπορούσα να δώσω ένα Ιρλανδικό παράδειγμα λύση, είναι ότι παρά το τεράστιο έλλειμμα στη ζήτηση, διότι όσα ε, επιδόματα κοινωνικής προστασίας παίρνουν ε, οι άνθρωποι από το σύστημά μας, αυτά επιζητούμε να, να δαπανώνται κιόλα εντός της χώρας, στα καταστήματά μας, στο εμπόριο της Ιρλανδίας. Τώρα για τους νέους. Είναι συνολικότερο το φαινόμενο της ανεργίας και πλήττει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όμως ειδικότερα για τους νέους, εδώ υπάρχει μια πρόσθετη πίεση Εξ όσων γνωρίζουμε από τις στατιστικές μελέτες, η ανεργία σε πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής φαίνεται στους νέους να είναι διπλάσια από ό,τι σε μεγαλύτερες ηλικίε. Διότι οι νεοαθιχθέντες στην αγορά εργασίας είναι εκείνοι που δυσκολεύονται περισσότερο. Αυτό είναι και το τοπίο εντό του οποίου γίνεται τόσο σημαντικό αυτό το κονδύλι της εγγύηση για τους νέους. Εδώ θέλουμε να τους ε, στηρίξουμε την εμπιστοσύνη τους ε, σε εμάς και έχουν τόσο καλή εκπαίδευση που είναι αδικία να μην βρίσκουν δουλειά. Θα πρέπει να έχουν λοιπόν ευκαιρίες και για εργασία και για περαιτέρω εκπαίδευση. Η πρώτη θέση εργασίας είναι άκρος σημαντική για νέους που μπορεί να είναι και θύματα κοινωνικού αποκλεισμού και για επιπλέον άλλους λόγους, αλλά σίγουρα ένας τρόπος ένταξης η έβρεση εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας θα, προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και το θέμα αυτό. Είναι προτεραιότητα για το Συμβούλιο ε, και νομίζω ότι αν βρούμε ένα κοινό πλαίσιο όπου θα συνεννοηθούμε και με το Κοινοβούλιο, θα είναι σημαντικό ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας οι άνθρωποι στην Ευρώπη, ιδίω οι νέοι. Και για να επιστρέψουν στην παρατήρηση του κυρίου Σέρκας, έτσι θα έχουν και χρήματα στα χέρια του για να τα δαπανίσουν και θα στηρίξει αυτό και την οικονομία. Σημαντικό είναι ο ρόλο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίω των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ θα θέλαμε και περισσότερε ευκαιρίε για του νέου, αλλά και του μεγαλύτερου, να μπορούν να ξεκινήσουν δικέ του επιχειρηματικέ προσπάθειες. Να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα εφόδια για να το κάνουν αυτό. Γιατί το πνεύμα του επιχειρήν είναι σημαντικό μέρο τη Ευρωπαϊκή ανάκαμψη συνολικά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα για την αυτόματη σταθεροποίηση, τους παράγοντες σταθεροποίησης. Για αυτούς τους λόγους ε, έγιναν αυτές οι παρατηρήσεις από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου επιμείναμε περισσότερο σε αυτή την επιλογή παρά στην μέθοδο ανοιχτού συντονισμού διότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή, αυτός ο αυτοματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτιμήσαμε λοιπόν την εγγύηση για τους νέους. Θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για να λειτουργήσει ακριβώς σε ευρωπαϊκή κλίμακα και να εξαλειφθούν οι μακροοικονομικές ελλείψεις ισορροπίας που γνωρίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω ότι ότι αυτά ξεπερνούν λίγο το πλαίσιο των διπραγματεύσεων, των δικών σα αρμοδιοτήτων, των δικού σα χαρτοφυλακίου στο άτυπο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, αλλά είναι σημαντική διάσταση που πρέπει να έχουμε κατά νου για τι επικείμενε αποφάσει του Ευρωκοινοβουλίου. Ο κύριο Κάνων, γιατί σα τέθηκαν ερωτήσει για το δυσχερέστατο θέμα του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε. να πω κάτι που προέκυψε από όλε τις ε, παρεμβάσεις. Υπάρχουν ε, ε, σημαντικά προβλήματα τόσο για τους άνεργους νέους όσο και για εκείνους που είναι μακροχρόνια άνεργοι. Αν δείτε λοιπόν τους στόχους, θεματικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο EFSF υπάρχουν κάποιες ελπίδες ότι αυτές οι προκλήσεις ε, θα αντιμετωπιστούν ε, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού. Η θεματική στόχη είναι η προαγωγή της απασχόλησης και η υποστήριξη της εργασίας, έρευνες ε, όσον αφορά τις δεξιότητες και την διαβιουμάθηση, προαγωγή, την ένταξη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και τέλος να προσφέρεται καλύτερη υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς και από τη δημόσια διοίκηση. Εμείς θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επενδύσεις στον τομέα αυτό ε, καθώς ε, αρχίζει να λαμβάνει ο κανονισμός αυτό στην τελική του μορφή. Πολύ καλά. Τέσσερις επόμενοι ομιλητές. Κλείνουμε εδώ τον κατάλογο ομιλητών, ναι. τσούτε. Νταρντέν, Ιασλοβιετσκά et ensuite le dernier bloc, ça sera και μετά τελευταία ομάδα. Εσάια Αρκίν. Εντάξει, μετά από τα ονόματα αυτά που μόλις ακούσατε, κλείνουμε τον κατάλογο των μιλητών. Ναι. Λίνκεβίτσε τούτη. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Πυρμηνίνκια, πριμάουσα νόριου παντιοκότη, δυσιαμ στριμ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω και τους τρεις Ιρλανδούς υπουργούς. Πράγματι, οι στόχοι σας είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Πιστεύω ότι η Ιρλανδία θα τα καταφέρει. Δεν είσαστε τίποτε πρωτάριδες, είναι η έβδομη φορά που αναλαμβάνετε την Προεδρία. Κάποιες ερωτήσεις τώρα. Ο Υπουργός ε, Μπέρτον Μα είπε ότι εξετάζεται την οδηγία κατά της διακριτική μεταχείρισης η Ιρλανδική Προεδρία. Τι προβλέψεις κάνετε για τα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις στον τομέα αυτό. Το όλο ζήτημα έχει, φαίνεται να έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεύτερη ερώτηση προ τον Υπουργό Μπέρτον. έχετε στα χέρια σας μια πολύ σοβαρή προτεραιότητα που αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και το τεράστιο αριθμό ανέργων. Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί ένα ε, έδαφος συνεννόησης προκειμένου να δοθεί στήριξη και σε όσους πλήττονται από τη φτώχεια. Διότι εδώ πραγματικά θα παίξουν σοβαρότατο ρόλο οι απόψεις των ίδιων των κρατών μελών. Και έπειτα για τον Υφυπουργό Κάναν και για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό το Ταμείο αυτό για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια πέτυχαν αρκετά στην χρήση του Ταμείου. Χάρη στη χρήση του Ταμείου. Κάποια άλλα όμως, κάποια άλλα πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξή του. Εσείς ποια συμβαστική λύση διαβλέπετε ως πιθανότερη. Και έπειτα έχω και μια ερώτηση για το πρόγραμμα Εράσμους. Πολύ σημαντικό και αυτό για τους νέους. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σε σχέση με την συνέχεια του προγράμματος Εράσμου στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Να θέσω ευθύ αμέσω τι ερωτήσει μου. Να σα ρωτήσω για την ανεργία μεταξύ των νέων. Στην Ιρλανδία, μια και το αναφέρατε. Ποια είναι η εξάπλωση της ανεργίας, σε ποιες κατηγορίες νέων αφορά περισσότερο στις ηλικίες 15 έως 30 ετών και ποια είναι η κατάσταση αυτής της ηλικία ομάδας είναι άνθρωποι που δεν σπουδάζουν, δεν δουλεύουν καν, δεν έχουν παροχή καμία μορφή εκπαίδευση. Τι μηχανισμού στήριξη προβλέπετε για του νέου, Νέου που μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν μια δική του επιχείρηση, μια δική του δουλειά. Και για το σύστημα τη εγγύηση για του νέου, αυτό που αναφέρατε στην ομιλία σα αρχικά. Τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, πιστεύετε, για να αλλάξει η κατάσταση, η θέση των νέων στην σημερινή αγορά εργασία. Μία λύση θα ήταν όντω αυτό το σύστημα εγγύηση. Όμω, μήπω ενέχει κινδύνου, μήπω η εισαγωγή ενό τέτοιου συστήματο ουσιαστικά ε, επιβαρύνει άλλε ομάδε τη κοινωνία μα. Νεαρέ μητέρε που θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασία και να ξαναδραστηριοποιηθούν. Λοιπόν, ίσως και 30 χρόνια αν κάτι έχω μάθει. Φρεντερίκ Νταρντέν και μετά ο επόμενο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ για όσα είπατε Χαίρομαι. Έχετε πιστεί ότι έχει προτεραιότητα αυτή η εγγύηση για τους νέους. Για μας είναι σημαντικό και επίσης για την προστιθέμενη αξία των κοινωνικών ταμείων όπως αυτό που προσφέρουν στους ασθενέστερους ε, σχετικά με την εγγύηση για την ηλικία και τα κράτη-μέλη στη ρύθμιση τους πρέπει να συμπεριλάβουν αυτόν τον όρο και τα μέσα μέσω ενό μέρους του κοινωνικού ταμείου είτε με ειδικό κονδύλι, ταμείο μάλλον ε, και σχετικά με την παγκοσμιοποίηση. Όλοι μας είμαστε πεισμένοι ότι χρειάζεται αυτό να διατηρηθεί αλλά ορισμένοι δεν είναι και το υπενθύμησε ένας από τους συναδέλφους σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε κανείς να καταλήξει κάπου σχετικά με αυτό και ακόμα χρειάζεται να είναι περισσότερο αποτελεσματικό με περισσότερους που θα απολαμβάνουν της βοήθειάς του και χρειάζεται βέβαια μέσα γι' αυτό και μήπως θα έπρεπε να προλαβαίνουμε αυτό αναφέρθηκε εδώ στη συζήτηση και στα πλέμα της έκθεσης Σύρκαζη για την αδιάρθρωση και για τη βοήθεια στα περισσότερα μειονεκτικά άτομα Μήπως θα έπρεπε με τους στόχους τους 2020 και της μάσκα της φτώχειας να συγκλίνουμε τους στόχους και να γίνει κάτι το συγκεκριμένο και μάλιστα στα γρήγορα και επίσης ολοκληρώνοντας έτσι σαν ε, τελικό συμπέρασμα όταν ακούω τα όσα λέτε και δεν με εκπλήσει Άλλωστε, τα πάντα εξαρτάται από τα πόσα χρήματα θα δοθούν και τα μέσα που θα δοθούν και το πολιετές πλαίσιο. Και εδώ να σας πω ότι εμείς εξαρτώμεθα από τα μέσα που θα μας δοθούν, χωρίς όμως να είμαι σίγουροι για τα μέσα που θα μας δοθούν. Εσείς θα πείσετε τους υπουργού οικονομικού σας και τους πρωθυπουργού σας ότι θα υπάρχουν αυτά τα μέσα, θα υπάρξουν αυτά τα μέσα. Είναι ήδη πεπισμένοι μάλλον. Ακούστε, μισό λεπτό και εσείς ζητήσατε λόγο, ναι, ναι θα σας σημειώσω, εντάξει, αν έχουμε το χρόνο, ε, κυρία Τζαχουδιέσκα, θα σας συμπεριλάβουμε και εσάς. Μάλλον όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω του ε, εκπροσώπου τη Ιρλανδική Προεδρία. Παρουσιάζεται πολλού φιλοδοξού στόχου και εκπλήσωμαι, διότι πραγματικά εδώ και χρόνια δείχνει την υπευθυνότητά τη και τη φιλοδοξία τη συστηματικά η κοινωνία τη Ιρλανδία. Καλή επιτυχία λοιπόν στο δρόμο σας. Η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων νομίζω θα είναι μια από τις πετεραιότητε της Προεδρίας όπως είπατε. Ε, είναι μια οδηγία που προκαλεί κατακραυγές κάποιες φορές. Κάποιες διατάξεις θεωρούνται προβληματικές για κάποιες κοινωνικές ομάδες ή σε κάποιες χώρες. Ελπίζω να υπάρξει καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της Προεδρίας σας. Η Ιρλανδική Προεδρία ξεκίνησε δίνοντας έμφαση στις αποταμιεύσεις της εξοικονόμηση κονδυλίων και την ανάπτυξη. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις όποτε προκύπτει μια κρίση. Είναι λογικό ε, να προσέχει κανείς για να αντιμετωπίσει τα χειρότερα. Η δική μα όμω επιτροπή επικεντρώθηκε στι κοινωνικέ επενδύσει με μια έκθεσή τη. Και αυτή είναι πολύ σημαντική για το Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Προβλέπετε δράσει που θα προωθήσουν τι κοινωνικέ επενδύσει. Νομίζω ότι το πιο σοβαρό κεφάλαιο, το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει η Ευρώπη είναι οι ίδιοι πολίτε, οι άνθρωποι τη. Και αυτό σε καιρού κρίση είναι ζωτική σημασία. Επίση, αναφέρατε το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Προβλέπετε δράσει που να συμπληρώσουν αυτό το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πάλι το λόγο έχουν οι τρεις υπουργοί, ίσως να αλλάξουμε τη σειρά παρέμβασής τους. Να συμφωνείτε εσείς ε, κύριε Κάνον να ξεκινήσετε για να αλλάξουμε τη σειρά απαντήσεων τώρα. Να πω πάλι ότι υπήρξαν ε, παρατηρήσεις ε, σε όλα τα σχόλια. Όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, εμεί στην Ιρλανδία ε, συγκεντρώσαμε αρκετή εμπειρία σχετικά με τη χρήση αυτού του Ταμείου. Έχει ωφελήσει πάρα πολλού ανθρώπους. Τους βοήθησε να βρουν κάποια θέση εργασία, να μπορέσουν να επανέλθουν στην εργασία. Έτσι λοιπόν το Ταμείο παγκοσμιοποίηση ήταν πολύ ε, σημαντικό στην Ιρλανδία. Μερικοί μπόρεσαν να επανέλθουν άμεσα, άλλοι μπόρεσαν να αποκτήσουν ε, δεξιότητες μέσα από την ε, περαιτέρω κατάρτιση και αρκετοί από αυτούς άνοιξαν τις δικές τους τις επιχειρήσεις μετά από την εμπειρία που συγκέντρωσαν σε προηγούμενες εργασίες. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως σε ε, σημαντικά κέντρα όπως τα call center που χάσανε και κλείσανε, κλείσανε και χάσανε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Πράγματι, πολύ επιτυχημένο ε, το Ταμείο αυτό. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον του Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν χώρε ε, που το στηρίζουν και άλλοι πάλι που λένε ότι δεν έχει καμία σημασία. Ε, Προφανώ, αυτό σχετίζεται άμεσα με τι συζητήσει που γίνονται για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης ε, πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης σε σχέση με το EFSF ε, γιατί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης τελικά απέδειξε ότι είναι πολύ καλύτερα σε θέση να ανταποκριθεί σε μαζικές ε, απολύσεις πολύ περισσότερο από το EFSF και κυρίως όταν τίγεται μια τοπική οικονομία. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ότι το κλείσιμο επιχειρήσεων θίγει περιοχές πλήττονται περιοχές επανειλημμένα που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτή την ξαφνική καταστροφή. Όσον αφορά τώρα του να επεκταθεί το Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να αντιμετωπίζει και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Αυτό δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ελέγχεται αυστηρά ο στόχος του Ταμείου έτσι ώστε να εστιάζεται περισσότερο σε πραγματικές ε, απολύσεις όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει μερίδια από την αγορά ε, στην περίπτωση αυτή μπορεί να βοηθήσει το Ταμείο με καλύτερη κατάρτιση των υπαλλήλων για να επανέλθουν στην εργασία. Το ESF, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μπορεί και αυτό ε, να ε, βοηθήσει στην ε, για να προκύψει πιο εύκολα αναδιάρθρωση στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Με οποιαδήποτε σειρά και σας βάλω, εσείς κυρία μου θα είστε πάντα στη μέση. Ήταν ε, πολλαπλά τα ερωτήματα, αλλά... Ήταν πολλαπλά τα αλλά εγγύηση για τους νέους και η ερώτηση που έγινε από την Τζοάννα για τη χρηματοδότηση αυτού του ταμείου για τις, τις για τους νέους. Η σύσταση προβλέπει χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Ταμείο να ε, αξιοποιηθεί για τη δημιουργία των συστημάτων εγγύησης για τους νέους. Όμως, όπως είπε και ο κ. Σάντορ, το συνολικό, η συνολική προκοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου και των άλλων Ευρωπαϊκών Ταμείων θα κρυθούν και από τι διαπραγματεύσει και την πορεία που θα πάρουν οι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων τα κάτι μέλη θα πρέπει να θέσουν προτεραιότητες και να θέσουν και ως προτεραιότητα αυτή την εγγύηση για τους νέους. Τέθηκε μια άλλη ερώτηση για τα επίπεδα ανεργία. στην Ιρλανδία, επειδή σε αυτήν αναφερθήκατε. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή φτάνει, το ποσοστό φτάνει το 14,6% και το ποσοστό των νέων είναι σχεδόν διπλάσιο. Αλλά όπω και στα περισσότερα μέλη νομίζω οι νέοι έχουν υψηλή εκπαίδευση και μεγάλη ε, κατάρτιση. Οι νέοι αυτοί λοιπόν μένουν άνεργοι συνήθως για μικρότερα διαστήματα από ότι νέοι που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Δεν νομίζω η Ιρλανδική περίπτωση να διαφέρει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως λόγω της οικονομικής κατάρρευσης στην Ιρλανδία, όπως και πολλοί από εσά ανησυχούμε ιδιαιτέρως για τους νέους. Νέους άντρε, οι οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο πριν καν ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο σκοπός λοιπόν δεν είναι απλώς να γεμίσουν τα ταμεία για την εγγύηση των νέων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην Ιρλανδία. Έχουμε δαπανίσει μεγάλο ποσό των πόρων του κοινωνικού ταμείου που ακόμη στέλνει προς την Ιρλανδία προκειμένου να καλύψουμε τους νέους. Μίλησα και για που χάνουν τη δουλειά του, ξαφνικά, αλλά θα πρέπει να έχουν και δυνατότητε να εκπαιδευτούν εκ νέου. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε πρωτοβουλίε στο Υπουργείο στο Υπουργείο μα για κάποιου που χάνουν τη δουλειά του από τον τομέα των κατασκευαστικών, μηχανικού λόγω χάρη. πρέπει και εκείνοι να μπορέσουν να εκπαιδευτούν περισσότερο. Ενδεχομένως σε νέες τεχνολογίες, στην πληροφορική. Εκεί μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις σε συγκεκριμένε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και εταιρείε. Υπάρχουν λοιπόν και θετικές δυνατότητες ε, μέσα από την κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα για τους παράγοντες σταθεροποίηση, όπως τους ανέφερε η Πρόεδρος. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασία, διότι σε μια περίοδο ύφεση θα πρέπει κανείς να κάνει εξοικονόμηση προκειμένου να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης, ιδίως για τους πλέον μειονεκτούντες. Και πάλι όμως, εξετάζοντας τις Ιρλανδικές στατιστικές στο ε, πλαίσιο της κρίσης και σε σχέση με τις μητέρες, που, τις μόνες μητέρες η, το ποσοστό αυτό ε, στην Ιρλανδία φτάνει το 61% σε σχέση με τους πόρους που δαπανήθηκαν για τον μετριασμό ακριβώς των συνεπειών της κρίσης και την ε, φτώχεια, το ενδεχόμενο της φτώχειας. Τα περισσότερα κατημέλη το ποσοστό αυτό είναι το μισό και σωστά ανέφερε η πρόεδρος τους παράγοντες σταθεροποίησης, διότι το έλλειμμα της ζήτησης έχει τεράστιο αντίκτυπο αλλάζουν οι ανάγκες και η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών στις εταιρείες της χώρας και βεβαίως υπάρχει και τεράστια επίδραση στα ποσοστά φτώχειας και άλλων δικτών κοινωνικής ένταξης. Ως προς το θέμα των νέων που ξεκινούν δικές τους δουλειές, το αποτελεί μέρος οποιοδήποτε προγράμματος για τους νέους, πιστεύω. Στην Ιρλανδία στηρίζουμε ανθρώπους κάθε ηλικία να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις ε, και βεβαίως εδώ έχουμε μια δυνατότητα νέων θέσεων απασχόλησης. Και είναι πολλοί νέοι που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν δικές τους πρωτοβουλίες, δικές τους προσπάθειες του επιχειρήν. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ίσως μια στιγμή δεν δει τα πράγματα ακριβώ, αλλά για την στρατηγική υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασία. Εκεί είμαστε ιδιαίτερα κινητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι. Περιμένετε μια πρωτοβουλία τη Επιτροπή για τη στρατηγική αυτή, αλλά δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να υπάρξει και ένα κάποιο χώρο για μια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Προεδρία, ώστε να θέσει επιτάπητο την ανέωση αυτή τη στρατηγική για υγεία και ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για την κυρία Μπλινκεβιτσιούτα. Μιλήσατε για την οδηγία κατά της διακριτικής μεταχείρισης. Είναι σημαντική οδηγία αυτή. Ε, όντως ασχολείται με την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες και εδώ θέλουμε να επιτελέσουμε πρόοδο. πρόοδο συγγνώμη. Εδώ βεβαίως ε, υπάρχουν προβλήματα, ιδίως λόγω της νομικής ασφάλειας που επιζητούμε και σε σχέση με το τι ισχύει από την η κυρία Ζαγοβλέσκα μίλησε για την οδηγία απόσπαση εργαζομένων. Ξέρω ότι εργάζεται επισταμένο ω εισηγήτρια για το θέμα αυτό και είναι και για μα προτεραιότητα. Θα καλωσορίσουμε την θέση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Ακόμη και αν δυσκολευτούμε να βρούμε κάποια συμβαστική λύση, κάτι θα πετύχουμε τι διαπραγματεύσει Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί ένα κοινό πεδίο συνεννόησης για τα δύο εκκρεμή σημεία. Θα τα συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο. Μιλήσατε για τη σημασία των κοινωνικών επενδύσεων και των σχετικών πρωτοβουλειών. Εδώ καλωσορίζω όπως για τις κοινωνικές αλλαγές και την καινοτομία, νέα εργαλεία που στηρίζουν τα μικροοικονομικά, την κινητικότητα, τη χρηματοδότηση νέων τομέων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ε, στήριξη των ε, υποδομών από τα κράτη-μέλη. Μιλήσατε και για την υγεία και την ασφάλεια και τη σχετική στρατηγική. Εδώ όντως θα αναλάβουμε στρατηγικές πρωτοβουλίες όταν υπάρξει σαφές τοπίο για το θέμα αυτό και σαφείς πρωτοβουλίες. Πρόεδρος. Ίσως πρέπει να βοηθήσουμε την Επιτροπή στο σημείο αυτό. Λοιπόν, τελευταία ομάδα ομιλητών. Καστέλο και επόμενος μετά. Καστέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις υπουργούς που ήρθαν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που άκουσα ότι η Ιρλανδική Προεδρία ε, στα προγράμματά της θέλει να συμπεριλάβει μια ουσιαστική κοινωνική διάσταση και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί έχουμε 16 ε, εκατομμύρια που κινδυνεύουν από φτώχεια και 40 περίπου εκατομμύρια που υποφέρουν από στέρηση αγαθών και δικαιωμάτων. Όπως είπε και ο Υπουργό, ε, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική συμπερίληψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Εμεί έχουμε έρθει σε επαφή με πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο, ε, γαλλικέ, βελγικέ οργανώσει και κάποιε γερμανικέ και Ιρλανδικέ ΜΚΟ. Και όλοι λοιπόν μα είπαν ότι το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό για την εξάλληψη τη φτώχειας ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι ε, παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται και άλλα μέτρα πολιτικής ε, για να περιοριστεί η ανέχεια. Καλωσορίζω λοιπόν αυτά που είπε η Ιρλανδική Προεδρία για τις εγγύησεις για τους νέους και προσβλέπω να συνεργαστώ μαζί σας. Και μια τελική ερώτηση που έχει σχέση με τις εγγύησει για τους νέους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το προβάλλουμε στο πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα και για τη μαθητεία είναι σημαντικό οι ε, νέοι που περνάνε από ε, τέτοια προγράμματα μαθητής να μην είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ε, υπόθηκε αυτό προηγουμένως ότι το Ταμείο για τους έχονες μεγαλύτερη ανάγκη είναι καθοριστική σημασία και θέλουμε να ενισχυθεί. Η Ευχαριστώ πολύ. Απ' έξω έχουμε μια μεγάλη διαδήλωση που αφορά στην εφαρμογή της οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων. Και ερωτώ λοιπόν αυτό το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων. Ε, τι σημασία έχει για την Ιρλανδική Προεδρία. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Εδώ ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την εισαγωγή μιας ε, τέταρτης πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Εσείς αναφέρεστε πιστικά στη σημασία του αγώνα κατά της ανεργίας των νέων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και ερωτώ όσον αφορά αυτό τον τέταρτο άξονα, την τέταρτη αυτή διάσταση. Τι ακριβώς έχετε να πείτε επ' αυτής. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ απευθύνομαι ε, στον Υπουργό Τζον Μπέρτον. Είπατε, ε, αναφέρατε το επισητιστικό πρόγραμμα και ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο δεν υπάρχει ε, συμφωνία για το θέμα της επιστικής βοήθειας. Ορισμένα κράτη-μέλη λένε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό, αλλά εθνικό, εθνικής κοινωνικής πολιτικής. Και θέλω να ακούσω περισσότερα από αυτού. Κατόπιν, ένα άλλο ερώτημα με το πρόγραμμα επιστηστικής βοήθειας. Η διανομή των τροφίμων σε πολλά κρατημέλη γίνεται από ΜΚΟ και από την Εκκλησία. Αυτοί βοηθάνε πάρα πολύ και με το νέο λοιπόν πρόγραμμα ποια θα είναι η θέση που θα καταλάβουν γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται μόνο το να δώσει κανείς ένα σακί τρόφιμα, να υπάρχει και κάποια κοινωνική επαφή. Ποια θα είναι λοιπόν στο μέλλον η θέση των ΜΚΟ και της Εκκλησίας στο πλαίσιο αυτού του επισητιστικού προγράμματος. Μαχριάν Αρκή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους τρεις υπουργού και να τους ευχαριστήσω και για τη δουλειά τους. Με συγχωρείτε που δεν ήρθα νωρίτερα. Δεν ήταν δυνατόν. Απλώ κάποιε ερωτήσει για όλου σα. Για τον κύριο Κάνον, μιλήσατε για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ όντω υπάρχει μια μειοψηφία που μπλοκάρει την εξέταση του θέματο. Εσεί, ω Ιρλανδική Προεδρία, πώ θα πείσετε του υπολείπου ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν με την πρόταση αυτή. Η πρόταση του Κοινοβουλίου νομίζω είναι μια καλή βάση για όσα θέλετε να κάνετε. Έχετε καινούργιε ιδέε όμω. Αυτή είναι η ερώτησή μου προ εσά. Στον Υπουργό Μπέρτον. Στην Υπουργό Μπέρτον, μάλλον. Αναφέρατε το πρόγραμμα για του μειονεκτούντε. Ε, και εσεί και άλλοι και τι συνάδελφοι. Κοίταξα τώρα το σχέδιο νόμων προτείνουν οι Βουλή των Λόρδων, η Bundestag. Λένε ότι ήταν πολύ καλά όταν υπήρχε επιστημιστική βοήθεια και σε σχέση με την ΚΑΠ αλλά τώρα δεν βλέπουν ότι κάτι τέτοιο είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αναλυθεί πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο. Ε, δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά εσείς πώς, πώς σκοπεύετε να ασχοληθείτε και με αυτές τις απόψεις, πώς θα τις καλύψετε. Είναι σημαντικό αν θέλουμε να πετύχει το πρόγραμμα. Και έπειτα για την εγγύηση για τους νέους. Πώς διαβλέπετε, και αυτό είναι περισσότερο Ιρλανδικού χαρακτήρα ερώτημα, πώς βλέπετε να συνδυαστεί αυτό με το Εθνικό Πρόγραμμα Μαθητιών και Ασκήσεων. Θα πετύχει και ένα σχόλιο για τις ανησυχητικές για τα ενισχυτικά ποσοστά ανεργίας. Μην ξεχνάμε εδώ πόσα υψηλά ποσοστά μεταναστών έχουμε. 70.000 μόνο ήρθαν πέρσι. Ε, λοιπόν, ε, πρέπει εδώ και την πολιτική μετανάστευση να την δούμε από κοινού. Η κυρία Ρέγνερ έθεσε εδώ μια ερώτηση, Υπουργέ Μπρέτον. Και πρέπει να δούμε όλα τα θέματα από κοινού. Το Συμβούλιο δεν φαίνεται να προχωράει με ταχύτητα στις διαπραγματεύσεις και έχουμε πολλές δυσκολίες. Εσείς τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για να προχωρήσουν όλοι οι άξονες ταυτόχρονα και για την απόσπαση των εργαζομένων και την οδηγία για την μη διακριτική μεταχείριση. Αυτά έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βίλτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εύχομαι στους τρεις υπουργούς πλήρη επιτυχία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτό το εξάμεινο και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς νομίζω ότι δεν προσέχουμε πως πρέπει τους νέους σε ηλικία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής για τον κύριο Μπρίτον Ρίτσαρντ ποια θα είναι η προτεραιότητά σας κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας ακριβώς για κάτι καλύτερο σε σχέση με τους μισθούς, γιατί είχαμε στο Κοινοβούλιο μια έκθεση. Εσείς πώς θα προωθήσετε το θέμα σχετικά με αυτό. Λοιπόν, πριν να πάρουν το λόγο και πάλι κύριοι Υπουργοί, να ζητήσω από τον Υπουργό κύριο Κάνον ε, για απαντήσει στο ερώτημα για τον ε, έρασμο. Έτσι, για να μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα και διαφορετικά να μας πείτε ποιος είναι ο αρμόδιος υπουργός. Ε, θα βοηθούσε την ε, Επιτροπή μας. και ίσως τον κύριο Μπρούτον να ρωτήσω το εξή, γιατί νομίζω θα είναι υπεύθυνο ο αρμόδιος. Εσείς πώς θα βοηθήσετε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για την οικονομική νομική Υπάρχει και μια κοινωνική πτυχή η οποία προστέθηκε εκεί με μια εντολή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο όμως και υπό την Κυπριακή Προεδρία μια σημαντική πρωτοβουλία με την επιστολή αυτή που στάλθηκε από τη μία επιτροπή στην ΕΚΟΦΗΝ πριν από τέλος της χρονιάς ώστε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό έτσι δυναμικά και να γίνει κάτι το ανάλογο και κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Παραμένει ανοιχτό το θέμα. Έχετε το λόγο πάλι και οι τρεις σας από τρία λεπτά και θα ξεκινήσουμε και πάλι από τον Υπουργό κύριο, Υφυπουργό κύριο Κάνον. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι το Εράσμος αφορά το συνάδελφο μου κύριο Κουίν. Είναι εκπαιδευτικό θέμα. Εγώ έτσι ξέρω, δεν ξέρω. Δεύτερον, ε, κυρία Χάκιν όσον αφορά την ερώτηση σας για το ε, Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση. Εγώ είμαι στεναρός υποστηρικτής αυτού του προγράμματος και όπως είπα προηγουμένως το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει άμεση σχέση και με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνει επίκαιρο το Ταμείο αυτό. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες προτεραιότητες πιεστικές. Και είναι σημαντικό οι χώρες οι οποίες έχουν επωφεληθεί όλα αυτά τα χρόνια από το πρόγραμμα προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση πρέπει να προβάλλουν ουσιαστικά επιχειρήματα, χειροπιαστές αποδείξεις για το τι ακριβώς προέκυψε με τα ωφέλη που απορρέουν από αυτό το ε, ταμείο. Όσοι λοιπόν υποστηρίζουν αυτό το ταμείο πρέπει να υψώσουν λιγάκι τη φωνή τους. Αλλά όπως σας είπα, σε τελική ανάλυση, ε, σε αυτές τις ε, συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, εκεί θα ληφθεί η απόφαση κατά πόσον θα συνεχίσει να υπάρχει το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ή όχι θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε κάποια θέματα που έχουν σχέση με αυτά που είπαν οι Κάστελο Σασέρ και Χάρκιν σε σχέση με τη βοήθεια που παρέχεται σε ε, άτομα που απειλούνται από εξαιρετική ανέχεια, ιδιαίτερα μειονεκτούντες. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση δική σας και του Κοινοβουλίου γενικότερα θα είναι πολύ σημαντική οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, κρατικοί φορείς ε, έχουν ε, εξετάσει το θέμα και στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θέλω όμως να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την σημασία που έχει αποδώσει το ΕΚΟΦΗΝ παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι δεσμευμένη να αντιμετωπίζει την ανέχεια τους πένιτες και αυτό αναφέρεται και στους στόχους του 2020 ότι πρέπει να μειωθεί ο ρυθμός των ανθρώπων αυτών. Μιλάμε βέβαια για άτομα μεμονωμένα, οικογένειες και παιδιά. Το ταμείο το οποίο θα συσταθεί με τον νέο κανονισμό, εκεί πρέπει να διασφαλίσουμε να μην υπάρχει χάσμα ανάμεσα στην αντίδραση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για αυτούς που όλους μας, ε, μας ενδιαφέρουν και την πραγματικότητα. Ο στόχος της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι να καταστήσει δυνατή την υλοποίηση αυτού του Ταμείου από τον Ιανουάριο του 2014. Και βεβαίως η πρικοδότηση του Ταμείου εξαρτάται από την επιτυχία ή μη των διαπραγματεύσεων για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, είπατε ότι υπάρχει προηγούμενο στο Bundestag και στη Βουλή των Λόρδων. Εδώ ακολουθεί το πρόγραμμα γεωργίας που προϋπήρξε. Ε, θέλω όμως να πιστεύω ότι εδώ δεν θα πρόκειται μόνο για τα τρόφιμα, γιατί σε πάρα πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και κυρίως είναι εκείνες που κανείς δεν εργάζεται στην οικογένεια και όπου ακόμα και ε, τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επανέλθουν στην απασχόληση, κυρίως αυτούς που δεν έχουν εργασία. Εμάς στην Ιλλανδία μας απασχολούν ιδιαίτερα τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς να έχουν φάει σωστό πρωινό, που δεν μπορούν να φάνε ένα ζεστό φαΐ όταν ξεκινάνε την ημέρα τους και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά τα παιδιά θέλουμε να βοηθήσουμε και αυτές τις οικογένειες. Ίσως ε, μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο με ΜΚΟ που ενδιαφέρονται όχι απλά για τα τρόφιμα αλλά γενικότερα για τη διατροφή. Και αν το καταφέρουμε αυτό, ε, βεβαίως ε, αυτό ε, θα εξαρτηθεί και από την συνεργασία με τις ΜΚΟ και με άλλους φορείς. Σας λέω, προσβλέπουμε στην έκθεση e Όσον αφορά τώρα στην εγγύηση για τους νέους και ε, ε, την πρακτική εξάσκηση των μαθητευομένων. Υπάρχει στην Ιρλανδία ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, το οποίο ξεκίνησε με μια, πληροφορία, με μια πρωτοβουλία που βασίστηκε στο διαδίκτυο. Πολλοί ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα αλλά το μάλλον να σε ενημερώσω ότι το 50% που ολοκλήρωσαν αυτά τα μαθήματα, τα, τους κύκλους πρακτικής εξάσκησης, κατόπιν ε, βρήκαν δουλειά. Υπάρχουν παραδείγματα όπως η Γερμανία, η Φινλανδία, η Αυστρία. Ε, έχουν πολύ καλή εμπειρία όλη αυτή στη μαθητεία και ίσως η Ιρλανδία μπορεί να μάθει και να προσφέρει νέες ευκαιρίες, ε, ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους για να βρουν θέση εργασίας. Πρόεδρος, από την απάντησή σας συνάγω ότι το θέμα των τροφίμων και γενικότερα της διατροφής ε, παραμένει το επίκεντρο του προγράμματος. Ακόμα και αν είπατε ότι και αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, τα παιδιά που είναι σχολείο σε κάποια φάση να έχουν ε, σωστή διατροφή. Θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία να το ξαναστήσουμε στο πλαίσιο της σχετικής έκθεσης. Ο κύριος... Ε, ο επόμενος ομιλητής ε, για τρια τέσσερα. λεπτά. Ε, τέθησαν κάποια θέματα. Το πολύ λεπτό θέμα της απόσπασης των εργαζομένων. Και δείχνει το θέμα αυτό ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα κινητικότητας, να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται και στο δικαίωμα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτή την, την ισορροπία επιζητούμε. Επίσης, ε, η Μάρια Χάρκιν έφτιαξε το θέμα της κοινωνικής αλλαγής και της καινοτομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ πρόκειται για τον τέταρτο πυλώνα, ε, που δεν το στηρίζει όμως ε, το Συμβουλίο. Λέει υπάρχουν τρία κεφάλαια και όχι τέσσερα. Κατά την άποψή μου, τον επόμενο μήνα θα πρέπει να ξεκινήσει τριμερή συζήτηση για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να εξευρεθεί συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πρόκληση για την Προεδρία και για τις ε, τριμερείς ε, συναντήσεις. Θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τις ε, διαφορές. Εσείς κυρία Πρόεδρε, τίξατε το θέμα της κοινωνικής διάστασης που θα συμπεριλάβουμε στις συζητήσεις μας. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος στο νέο χάρτη που θα εξεταστεί κατά διάρκεια του εξαμήνου η ΕΠΣΚΟ θα έχει τη δυνατότητα να εξτάσει όλα αυτά τα θέματα ε, που θα επηρεάσουν την κοινωνική προστασία και πάρα πολλά άλλα. Και επίσης θα υπάρξει και η ε, παρουσίαση των απόψεων ε, στο ΕΚΟΦΗΝ. Ελπίζω λοιπόν ότι όλα αυτά να εξαστούν καλύτερα λόγω του ότι είναι πολύ σημαντικά. Σημείωσα βέβαια αυτά που είπε η κυρία Φοντανιέ που έχει μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη να τη λάβουμε υπόψη μας για να έχουμε μια πιο σφαιρική συζήτηση επί του θέματος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ε, απαντήσεις σας. Εγώ σας εύχομαι επιτυχημένη Ιρλανδική Προεδρία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στις ε, διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδική Προεδρία αποκομίσαμε θετικά θετικές εντυπώσεις. Ε, συνεχίζεται βέβαια ε, η τριμερή συνάντηση, καλό το χρονοδιάγραμμα, καλά τα συμπεράσματα που εξάγονται, δύσκολα βέβαια και με μεγάλη μας χαρά να σας δούμε πρώτα στο Συμβούλιο Απασχόλησης, ε, Κοινωνικής Πολιτικής κτλ, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ και στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ και όπως είπα και προηγουμένως θα υπάρξει συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας όταν θα έρθουμε να σας επισκεφτούμε στο Δουβλίνο. Και τώρα με μεγάλη χαρά να προσκαλέσω όλους σας σε μία μικρή δεξίωση για τη νέα χρονιά. Και ελπίζω να Υψώσουμε όλοι τα ποτήρια μας ε, εκφράζοντας ε, τις ίδιες ευχές. Ε, ξαναρχίζουμε στις 3.